Okay, colleagues, we are few, but... Uh, λοιπόν, συνάδελφοι, λίγοι και καλοί είμαστε. Τι να κάνουμε. Νομίζω. With travel. Δευτέρα απόγευμα είναι πάντα μια ώρα δύσκολη, διότι ταξιδεύουμε και συγκεκριμένη Δευτέρα ακόμα πιο δύσκολη από άλλες Δευτέρες. Είναι πολλά τα θέματα και πολύ φορτωμένη σήμερα η μερίσια διάταξη. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε λοιπόν. Ε, σημείο πρώτο, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μπορούμε να την εκρίνουμε όπως έχει. Δεν έχει ζητήσει κανένας καμία αλλαγή. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερο, ανακοινώσει τη Προέδρου. Δεν έχω εγώ ανακοινώσει αυτή τη στιγμή. Θέλω να σα πω μόνο ότι η τελευταία μα σε πριν τι εννέε διακοπέ και σε όσου δεν ξαναδώ, εύχομαι καλέ διακοπέ. Αν είστε μόνο για τα δύο πρώτα θέματα ε, εδώ, εμείς είμαστε μέχρι τις 6.30 αύριο το απόγευμα. Θα σας πω πότε θα έρθουν και ποιοι θα έρθουν στην Επιτροπή μας. Σημείο τρίτο, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 23ης και 24ης Μαΐου είναι ε, στους φακέλους σας. Αν έχετε σχόλια, δηλώστε το στην γραμματεία πριν το τέλος της ε, Επιτροπής, αλλιώς θα τα εγκρίνουμε. Τέσσερα. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις των συντονιστών, τα πρακτικά της 21ης Ιουνίου και πάλι. Αν έχετε σχόλια στη γραμματεία, αλλιώς θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά και αποφάσεις που εγκρίθηκαν καθώς και οι συστάσεις. Πέντε. Ανακοινώσεις Επιτροπής. Η, η Καθλίν με είναι παρούσα. Έχουμε και Γενική Διευθύντρια. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα σχόλια. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την ΤΕΦΚΟ δεν έχουμε καμία ανακοίνωση. Δεν ξέρω από την άλλη Γενική Διεύθυνση, εμείς πάντως όχι. Έχουμε το Γενικό Διευθυντή ΤΕΦΚΟ εδώ παρόντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ε, όλα αυτά τα χρόνια μαθαίνω ότι είναι η τελευταία σας συνεδρίαση. Αύριο θα είστε παρούσα γιατί έχουμε και ερώτηση. Ευχαριστώ. Καλή τύχη. Congratulations on your move για, για τη, τα υπερπόντια εδάφη και τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Σημείο 6, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη μετανάστευση. Με άλλα λόγια, είναι οι νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση και την κρίση αυτή μακροπρόθεσμα. Όχι τώρα το άμεσο προσφυγικό από τη Συρία, αλλά γενικότερα. η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συνεργαστεί κυρίω με χώρε τη Αφρική για να αντιμετωπιστούν ζητήματα τη μετανάστευση. Ο Στεφάνο Μασεβίση, Γενικό Διευθυντή ΤΕΦΚΟ, είναι παρόν εδώ. Για πρώτη φορά έρχεται εδώ σε συνεδρίαση τη επιτροπή μα. Στο παρελθόν ε, βέβαια είχε έρθει σε δύο ακρόασει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε μια νέα ανακοίνωση λοιπόν στις 7 Ιουνίου και βασικό στοιχείο αυτής είναι η ιδέα ε, του συμφώνου ή των συμφώνων μετανάστευσης στην αρχή με πέντε χώρες στην Αφρική, σε Μεγάλη, Μάλι, Νίγηρα, Νιγηρία και Αιθιοπία. Και θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε λίγο τι σημαίνει αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης. Γιατί ξέρουμε ότι η ανακοίνωση ε, προβλέπει και χρήματα, ένα δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον. Δηλαδή, 500 εκατομμύρια θα κοινοποιήσει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά λέει τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βάλουν ισόποσο. Ε, το συζητήσαμε αυτό με την κυρία Μογκερίνη. Υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει από πλευρά ε, κρατών μελών και κατά πόσο θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγάζει κάποια χρήματα, τα κράτη πού θα τα βρουν. Και άλλα θέματα, όχι μόνο τη χρηματοδότηση, πό, δηλαδή θα τα βγάλετε από τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βοήθεια. Τι γίνεται με την υποβόσκουσα αιρεσιμότητα, γιατί το συζητήσαμε την Πέμπτη, κάπως το βλέπουμε να συνδέεται περισσότερο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και λιγότερο στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή χώρε που είναι πρόθυμε να ε, υποδεχτούν ξανά πρόσφυγε στο έδαφο του και το συνδέουμε με την αναπτυξιακή βοήθεια, γιατί δεν έχουμε πολύ καταλάβει τι εννοείται. Το έχω πει και στην Ολομέλεια. Στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής από τη συνθήκη είναι να μειωθεί η φτώχεια. η οποία είναι ο βασικός ε, ε, παράγων και η αιτία που οθεί τον κόσμο να φεύγει από τη χώρα του και να βγαίνει στην πρόσφυγια. Θα μας πείτε λοιπόν πώς ε, λειτουργούν αυτά τα σύμφωνα, είναι εύκολο ή όχι και ποιο είναι το επόμενο βήμα. Κατά τα άλλα θέλω να σας πω ότι κάνουμε κοινή έκθεση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης ε, στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ συνδυάζει όλες τις πολιτικές μας πώς αποκρινόμαστε σε ζητήματα της προσφυγικής κρίσης και μετανάστευσης. Δίας Ντεμέρα και ερίκε Γκερέρο είναι οι συνεισηγητές. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει το Σεπτέμβριο. Αυτά. Κύριε Γενική, έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ανταλλαγή απόψεων, για παροχή πληροφοριών εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα όσα κάνουμε. Χρειαζόμαστε σαφώς αυτό τον διοργανικό διάλογο. Διανύουμε μια δύσκολη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε προ τα έξω ότι όντω συνεργαζόμαστε καλά ω ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όντω πρόκειται για ανακοίνωση τη Επιτροπή τη 7η Ιουνίου. Μια ανακοίνωση που αποτελεί ένα νέο βήμα μπροστά μια νέα προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο, αλλά το μοντέλο δεν είναι τόσο καινούριο τελικά, γιατί η διασύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη μετανάστευση είναι μια διασύνδεση που ήδη υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια. Γιατί πολλές φορές, όπως είπατε, ο λόγος μετανάστευσης συνδέεται και με τη φτώχεια, αλλά και με τη γενικότερη αστάθεια, αλλά ακόμα και με τις κλιματικές αλλαγές. Η διασύνδεση λοιπόν αυτή δεν είναι νέο φαινόμενο. Και θα πρέπει βέβαια να δούμε ότι υπάρχουν και κάποιες κρίσεις οι οποίες δεν είναι νέες. Ήδη από τη δεκαετία του 90 έχουμε κρίση στα Δυτικά Βαλκάνια και ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 2000 έχουμε μεταναστευτικές ροές που ξεκίνησαν τότε. Βασιζόμαστε λοιπόν σε ένα φαινόμενο το οποίο έχουμε εντοπίσει τα τελευταία χρόνια και σε κρίσεις που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια. Και στο παρελθόν δημιουργήσαμε και κάποιε διαδικασίε, όπω τη διαδικασία του Ραμπάτ και ο πρώτο πυλώνα για τη μετανάστευση και την απασχόληση στην πρώτη κοινή στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική ήδη μιλούσε για τη διασύνδεση αυτή. Πάντω, ανάπτυξη και μετανάστευση είναι δύο παράγοντε που έπρεπε να διασυνδεθούν. Σίγουρα αυτό δεν ήταν πολύ εύκολο. Έγινε μια πολύ μακρά συζήτηση όσον αφορά για παράδειγμα την ε, διαρροή εγκεφάλων. Δεν επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ στο ζήτημα των εμβασμάτων Έπρεπε επίσης να δούμε πώς θα καταφέρναμε να αποφεληθούμε από αναπτυξιακής πλευράς όσον αφορά το φαινόμενο της μετανάστευσης. Επομένως, ε, δεν μιλάμε για κάποιο νέο φαινόμενο, για κάποια νέα προσέγγιση, απλώς συνειδητοποιούμε σήμερα περισσότερο από ποτέ ότι θα πρέπει να συγκεράσουμε και να συνδυάσουμε τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Δεύτερον, τι άλλαξε τα ίδια τα μοντέλα της μετανάστευσης, οι ίδιες οι μορφές μετανάστευσης. Όχι μόνο έχουμε περισσότερα εκτοπισμένα άτομα, 65 εκατομμύρια παγκοσμίω, αλλά επίσης ο αριθμός των μεταναστών σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα 250 εκατομμύρια είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται περισσότερο από τον νότο προς τον νότο. Και Ακόμα και όταν ε, ασχολούμουν περισσότερο με τι εσωτερικέ υποθέσει στο παρελθόν, είχα πει ότι θα έπρεπε να συνδυάσουμε το ζήτημα τη μετανάστευση με το γενικότερο ζήτημα τη κινητικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε μόνο στα βαθύτερα αίτια, στα κίνητρα, αν θέλετε, τη μετανάστευση, αλλά στο γεγονό ότι οι άνθρωποι έχουν τα μέσα πλέον για να κινούνται περισσότερο. Και κατά τρίτο λόγο, αυτό το βλέπουμε και στο ότι ε, παλαιότερα οι ε, στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν αναφέρονταν στη μετανάστευση, ενώ τώρα το κάνουν. και βλέπουμε ότι το κάνουν αυτό όχι μόνο επειδή η μετανάστευση συνδέεται με το ζήτημα της κινητικότητας, αλλά επειδή έχουμε και κάποιες νέες διατυπώσεις όσον αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι στόχοι είναι πλέον πιο γενικοί, πιο σφαιρικοί. Επομένως, η μετανάστευση και η κινητικότητα αποτυπώνται πλέον καλύτερα στο θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030. Και είπαμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε κανέναν εκτός, ότι θα πρέπει να είναι στόχοι οι οποίοι θα απευθύνονται σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτά λοιπόν προσπαθήσαμε λοιπόν να εντάξουμε όπως είπατε εσείς και την αναπτυξιακή βοήθεια και υπάρχουν επίσης και πολλές διαφορετικές μορφές όσον αφορά το φαινόμενο αυτό. Σαφώς λοιπόν ξεκινούμε από την κρίση αυτή, αλλά δεν ανταποκρινόμαστε μόνο στην κρίση αυτή. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφερόμαστε σε διάφορα σχέδια τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε μια πολιτική όσο δυνατόν πιο σφαιρική. Ο πρώτος μας στόχος μας, ο πιο βραχυπρόθεσμος στόχος μας, θα θέλετε, είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Γιατί βέβαια καταλαβαίνετε ότι Όλοι οι πολίτε, όλοι οι μετανάστε κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή, διακινδυνεύουν τη ζωή του. Βλέπετε πώ έχουν τα πράγματα στην κεντρική Μεσόγειο, καθώ επίση και στην Ανατολική με την Εστευτική Οδό. Ο πρώτο μα λοιπόν στόχος στόχο να κάνουμε κάθε το δυνατό για να σώσουμε ζωέ. Δεύτερον και λίγο πιο μακροπρόθεσμα θέλουμε να δημιουργήσουμε καλύτερε συνέργειε ανάμεσα στην ανεπτυξιακή πολιτική και πραγματικέ επεμβάσει προκειμένου η δυνάμει μετανάστες ή πρόσφυγες να δούνε πώς έχουν τα πράγματα στη χώρα τους και ενδεχομένω να αναλογιστούν εναλλακτικέ λύσεις προτού αποφασίσουν να κινδυνεύσουν τη ζωή τους για να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερε θέσει απασχόληση ή να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι επιτόπου ή να αντιμετωπίσουμε τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή. Είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε να σώσουμε ανθρώπινε ζωέ και Κατά αυτόν τον τρόπο περνάμε στον πρώτο πυλώνα των συμφώνων αυτών, να καταφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να επέμβουμε, προκειμένου να βοηθήσουμε τις χώρες εταίρους να διαχειριστούν καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές. Και λέμε διαχείριση με την ροών και όχι συνόρων, γιατί θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να διαχειριστούν τα σύνορά τους, όπως ακριβώς το κάνουμε για να τις βοηθήσουμε να οικοδομήσουν ένα σωστό κράτος, αλλά το καλύτερο είναι να καταφέρουμε να τις βοηθήσουμε να αναχαιτήσουν και χειριστούν αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Μπορούμε να πλαισιώσουμε και να χειριστούμε αυτές τις μεταναστευτικές ροές, αν καταλάβουμε καλύτερα ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης ή και οι ευκαιρίες που υπάρχουν στις χώρες καταγωγής. Και είναι πολύ σημαντικό βραχυπρόθεσμα να έχουμε τα απαραίτητα θεσμικά όργανα, τα οποία θα είναι σε θέση να επιβάλλουν μια νομοθεσία, μια μεταναστευτική νομοθεσία. Να ακολουθηθούν δηλαδή συγκεκριμένε διαδικασίε όσον αφορά τη μετανάστευση και κατά αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πέφτουν στα χέρια των παράνομων διακινητών. Θέλουμε, θέλετε, περισσότερε νόμιμε οδού. Πράγμα το οποίο απαιτεί βέβαια από εμά να δούμε πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε πιο αξιόπιστη την διάθεση κάποιων συγκεκριμένων νόμιμων οδών. Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, η διαχείριση της σχετικής νομοθεσίας στις χώρες καταγωγής μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες ευκαιρίες για νόμιμη μετανάστευση και για την καταπολέμηση των διακινητών. Δεύτερον, και το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, στην εισαγωγή σας, τι μπορούμε να κάνουμε με τους επαναπροωθούμενους, με την επιστροφή. Ξέρετε ότι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία όσοι είναι παράτυποι μετανάστες πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες από τις οποίες προήλθανε. Πρόκειται για μια κοινοτική ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί με απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή στα άτομα όμω αυτά επιστρέφουν στη χώρα καταγωγή του, τι κάνουν εκεί πέρα. Θα του αφήσουμε μόνους του. Εγώ, όπω σα είπα, εργάστηκα στα πλαίσια των στερικών υποθέσεων ασχολήθηκα με το ζήτημα αυτό. Πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί απλώς επέστρεφαν στη χώρα τους, αλλά δεν υπήρχε καμία πλαισίωση από εκεί και πέρα. Βρισκόντουσαν, αν θέλετε, μόνοι τους στο μέσο του πουθενά. Και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζονται από τις κοινότητές τους ή από την οικογένειά τους σαν άνθρωποι οποίοι έχουν αποτύχει. Και Καταλαβαίνετε επίση ότι η όλη αποτυχία συνδέεται και με το γεγονό ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πλέον στο εξωτερικό και δεν μπορούν να στείλουν εμβάσματα στι οικογένειέ του. Πώ μπορούμε λοιπόν όχι μόνο να εγγυηθούμε την επιστροφή των ανθρώπων αυτών, αλλά και την αποτελεσματική επανεισδοχή και επανένταξη των ανθρώπων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και τι χώρε εταίρου και τους ανθρώπους αυτούς να επανενταχθούν στις κοινότητές τους, να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια μορφή απασχόλησης ή έστω μια μορφή κατάρτισης, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να καταφέρουν να ενταχθούν εκ νέου στην κοινωνία της χώρας καταγωγής τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε σαφώ την εσωτερική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τι επιστροφέ, αλλά δεν αρκεί να προωθούμε του ανθρώπου αυτού σε μία άλλη χώρα, χωρί στη συνέχεια να του βοηθούμε να ενταχθούν στην κοινωνία τη χώρα αυτή. Τρίτον, όλο και περισσότερο στι χώρε εταίρου μα, βλέπουμε ότι θα πρέπει να τι βοηθήσουμε ή να βοηθήσουμε μάλλον στι χώρε αυτέ, του ε, ανθρώπου αυτού οι οποίοι είναι απομονωμένοι πλέον, μπλοκαρισμένοι αν θέλετε σε μια χώρα, σε μια χώρα διέλευσης. Είτε επειδή έχουν ε, προσπαθήσει να ξεφύγουν από μια άλλη χώρα, είτε επειδή οι αρχές της χώρας διέλευσης ε, τους ε, έχουν σταματήσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο ή στον Νίγηρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τι μέτρα μπορούμε εμεί να πάρουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε του ανθρώπου αυτού, οι οποίοι βρίσκονται μπλοκαρισμένοι σε μια χώρα, στον Νίγηρα για παράδειγμα, ή στην Αιθιοπία. Ξέρετε ότι έχουμε μεγάλου καταβλισμού στο Ανατολικό Σουδάν, στη Σομαλία. Έχουμε πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται στου καταβλισμού αυτού και του οποίου θα πρέπει να του βοηθήσουμε. Για να βοηθήσουμε του ανθρώπου αυτού, πρέπει ουσιαστικά να βοηθήσουμε τι χώρε καταγωγή ή τι χώρε διέλευση, είτε να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να ενταχθούν στις τοπικές κοινωνίες ή να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους με τη βοήθεια της ΥΠΑ της Αρμοστίας των ΗΕ για τους πρόσφυγες. Αυτό πρέπει να γίνει με τον πιο αξιοπρεπή τρόπο και να τηρούνται πλήρως βέβαια τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης μέσω του πολιτικού διαλόγου να εγκρίνουμε και να εφαρμόσουμε μία νομοθεσία η οποία θα μπορεί να προστατεύει τους ανθρώπους αυτούς. Μία νομοθεσία που θα επιτρέπει στα άτομα αυτά τα οποία έχουν μια μορφή προστασίας να έχουν πρόσβαση στη συνέχεια στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να πλαισιώσουμε και να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά τα οποία βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Κάτι ακόμα πώς μπορούμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα του επίπεδου ασφαλείας σε συγκεκριμένες περιοχές. Ένα ζήτημα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη αυτή ανακοίνωση της 7ης Ιουνίου, αλλά το οποίο θα το λάβετε με τη μορφή νέας ανακοίνωσης, η ανακοίνωση CBSD. Δηλαδή, να καταφέρουμε να συνεργαστούμε με τις χώρες επιβολής του νόμου των κρατών αυτών, των χωρών εταίρων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις απειλές τρομοκρατίας. Αυτά εν γέννη όσον αφορά του βραχυπρόθεσμου στόχου μα. Ακριβώς όμως επειδή δεν ανταποκρινόμαστε μόνο βραχυπρόθεσμα και πολύ περιορισμένα σε μία κρίση, αλλά επειδή ακριβώ θέλουμε να ατενίσουμε, αν θέλετε, το μέλλον και λίγο πιο μακροπρόθεσμα, έχουμε προχωρήσει συγκεκριμένε προτάσει. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο δεν θα το αποκαλούσα καν φαινόμενο, είναι, αν θέλετε, μία τάση, μία διαφορετική τάση. Και βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν συγκεκριμένες δημογραφικές τάσεις, δημογραφικά χάσματα, ήδη και στην Ήπειρο της Αφρικής. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε ποια θα είναι η επίπτωση των κλιματικών αλλαγών, η αστάθεια που αυτές προκαλούν. Το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι λογικό να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες ζωής, ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα, τα οποία αντιστοιχούν ουσιαστικά στα βαθύτερα αυτά αίτια ή τα διαρθρωτικά αν θέλετε αίτια, τα οποία σπρώχνουν πάρα πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Δεν θέλουμε να εξαλείψουμε αναγκαστικά μόνο τα αίτια αυτά, αλλά να δημιουργήσουμε και περισσότερες ευκαιρίες για αυτούς τους ανθρώπους και να δώσουμε στα άτομα αυτά περισσότερες, αν θέλετε, νομικές εναλλακτικές οδούς για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια λοιπόν τη ανακοίνωσής μα, επικεντρωνόμαστε σε ένα βασικό στόχο, στην νεολαία, στους νέους οι οποίοι μας απασχολούν βέβαια στο παρόν, αλλά αποτελούν και το μέλλον της Αφρικανικής Υπήρου. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Αφρική. Αυτό θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μακροπρόθεσμα, θα θέλαμε να συζητήσουμε περισσότερο με τις χώρες αυτές και να επικεντρωθούμε περισσότερο στα πλαίσια του θεματολογίου της Αντίσα Μπέμπα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης επιτόπου, προκειμένου να δοθούν εναλλακτικέ στους ανθρώπους αυτούς και να παραμείνουν στη χώρα καταγωγής τους. Αυτά για την πολιτική. Τα μέσα που κινητοποιήσαμε είναι δύο είδων. Βραχυπρόθεσμα θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε το Trust Fund τουλάχιστον το τμήμα που συνδέεται με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Επίσης, αποφασίσαμε να προτείνουμε, γιατί τελικά τα κράτη-μέλη θα πάρουν την απόφαση, να κινητοποιήσουμε μισό δις ευρώ από ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε, Αναπτυξιακό Ταμείο, ούτως ώστε να έχουμε μια κρίσιμη μάζα κονδυλίων για αυτές τις πέντε χώρες που έχουμε ε, ορίσει ως προτεραιότητα. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Με αυτές τις πέντε θα δημιουργήσουμε μία δυναμική. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Διότι από τα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε συγκρίσιμες καταστάσεις. Είπαμε πως ε, ξεκάθαρα είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα και άρα όχι μόνο πρέπει να κινητοποιήσουμε τις ομολογουμένως ε, περιορισμένες δυνατότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, αλλά θα χρειαστεί, γιατί το λέμε συνέχεια πρέπει να τα κινητοποιήσουμε, αλλά ταυτόχρονα και το τονίζω σε αυτές τις πέντε χώρες και ξαναλέω θα ακολουθήσουν και άλλες θα πρέπει να συνεργαστούμε ούτως ώστε ο κοινό προγραμματισμό και η κοινή εφαρμογή να προωθηθούν. Κάποια κράτη-μέλη ήδη ε, έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτά τα κράτη-μέλη, όμως πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέρα από αυτά τα κράτη-μέλη, όλοι πρέπει να ανταποκριθούμε. Εάν δεν μπει φρέσκο χρήμα από τα, από τα κράτη-μέλη στο καταπίστευμα, γιατί ε, σίγουρα δεν είναι, δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό το Trust Fund, τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον να επιδιώξουμε ομαδοποίηση των κονδυλίων για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, γιατί είναι συλλογική δράση. Μακροπρόθεσμα τώρα, επειδή η βασική πρόσβαση είναι οι επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να φτιάξουμε ένα μέσο ε, που θα βασίζεται στα βιώματά μας. Με αυτά τα blending facilities για τις επενδύσεις, ε, για τις υποδομές, για την ενέργεια, ε, μείγμα επιδοτήσεων και δανείων δηλαδή, διότι ξαναλέω πρέπει να είναι νέο μέσο. Θα εμπνευστούμε από το blending, αλλά θα ε, καλύπτουμε τις ε, υπηρεσίες ε, για την εγγύηση των πιστώσεων. Αυτό δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, ούτως ώστε να υπάρχουν ισχυρότερες συνέργειες δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Μετά από την καθήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα καταθέσουμε κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο ε, μία νομοθετικού περιεχομένου πρόταση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ομαδοποιήσουμε διαφορε διάφορες δράσεις, όπως την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί ήδη δραστηριοποιείται σε αυτή την περιοχή. Θέλουμε συνέργειε. αυτό είναι το σύνθημα, θέλουμε μία κρίσιμη μάζα. Και για να πρικοδοτηθεί η προσπάθεια. Ό,τι έχουμε τώρα στα μέσα blending, 6 δις πάνω κάτω έχουμε, θα τα θέσουμε ε, στη διάθεση αυτού του προγράμματος για τις επενδύσεις. Θα προσθέσουμε και άλλα 100 εκατομμύρια. Και ξαναλέω τα κονδύλια, είναι ε, εθνικά κονδύλια. Θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη στο μέτρο των δυνατότητων να συνεισφέρουν. Μπορώ να πω ότι οι επενδύσεις για το blending μπορούμε να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα της τάξης του 10. Αυτά βλέπουμε στις μελέτες μας. Ξαναλέω, ομαδοποίηση κονδυλίων, προσθήκη επιπρόσθετων μέσων, blending συν ε, αυτά που μας δώσουν τα κράτη-μέλη επί 10. Αυτή θα είναι η δυνατότητά μας. Αυτά κάνουμε για να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Τελευταίο σημείο, Δεν ανταποκρινόμαστε έτσι σε μια τέτοια κρίση, αλλά θέλουμε να επιδιώξουμε ευρύτερη ευρωπαϊκή συνένεση. Πρέπει να ενσωματωθεί αυτό στην αναπτυξιακή μα πολιτική. Δεν, δεν κάνουμε κάτι εντελώ διαφορετικό. Πρέπει να πιστούμε ότι είναι τμήμα, ε, αναπόσπαστο κομμάτι τη αναπτυξιακή μα πολιτική. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε βάσει των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη ε, την μετανάστευση με πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο, με πολύ πιο ανοιχτό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν ω προ του στόχου τη χιλιετία δηλαδή και ήταν πολύ πιο κατακαιρματισμένο το κουτί εργαλείων που είχαμε τότε. Αυτό είναι το όραμά μας. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τώρα για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Θέλουμε βιώσιμα να δράσουμε. Ε, θα έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να το ξανασυζητήσουμε εάν να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Όλα δρομολογήθηκαν με αυτή την ανακοίνωση 7 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε συγκεκριμένα τι ε, αλλαγέ επισύρει αυτό. Πασχίζω να καταλάβω. Ε, σίγουρα οι συνάδελφοι θα έχουν ερωτήσει τώρα. Για να ακούσουμε κάποιες. Νόιζερ. Ντίβα. Νομπέρτ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και ε, της ανακοίνωσης αυτής και βέβαια παραμένουν πολλές ερωτήσεις ιδιαίτερα. Και πάλι από τον προπολογισμό παίρνετε κονδύλια για αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή σιγά σιγά έχουμε χάσει τον έλεγχο και δεν καταλαβαίνουμε πού πάνε τα χρήματα αυτά και πώς θα επιτύχετε αυτές τις συνέργειες που ζητάτε. Πραγματικά πάρα πολύ αφηρημένα τα βρίσκω αυτά, ειλικρινά σας το λέω. Μιλήσατε για βράχη πρόθεσμους στόχους, παράδειγμα, να σώζετε ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι αυτό το πράττουμε και στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αλλά δεν μπορούμε, ούτε το κάνουμε σε ένα τομέα, ε, ε, στην Αφρική μέχρι να φτάσουν στις ακτές της ε, Λιβύης, στη Μεσόγειο πού και πώς μπορούμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές στη Σαχάρα ή σε δύσκολα περάσματα ε, από την Αιθιοπία, Ερυθρέα, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Λιβύη, σε όλη αυτή τη διαδρομή πώς θα τους βοηθήσουμε και πώς θα σώσουμε ζωές. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πώς διαχειρίζεται κανείς μεταναστευτικές ροές. Αυτό εγώ το αντιλαμβάνομαι μόνο ως συνοριακούς ελέγχους. Δηλαδή στους ελέγχους τους βρίσκουμε και τους καταγράφουμε. Και από εκεί και πέρα τα ζητήματα και τα προβλήματα τα έχουν τα κράτη-μέλη. Εσείς είπατε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με τις χώρες εταίρους έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ε, φιλοξενούνται κοντά στις πατρίδες τους, για να το πω έτσι, και να έχουν μια προοπτική για τη ζωή τους. Εντάξει, αυτά μπορεί να είναι ήδη πραγματικότητες και δεδομένα, αλλά να τους δώσουμε εναλλακτικέ ε, που να αποτρέπουν τον κόσμο να φεύγει από την πατρίδα του. Όποιο για κάποιο λόγο φεύγει από τη χώρα του και προσπαθεί να σωθεί, μπορεί να βρει σωτηρία στη γειτονική χώρα, αλλά ε, μπορεί να χρειαστεί να πάει και παραπέρα. Μιλήσετε για διάφορες χώρες από τις πέντε αναφερθήκατε στον Ήγυρα και την Αιθιοπία ότι, ότι έχουν εκεί ε, φούσκες ε, ολόκληρες συγκεντρώνονται πάρα πολλοί πρόσφυγες σε χώρες πάρα πολύ φτωχές. Εγώ γνωρίζω από την Αιθιοπία ότι κάθε εβδομάδα έρχονται χίλιοι από την Ερυθρέα. 800.000 πρόσφυγες έχει αυτή τη στιγμή η Αιθιοπία στο έδαφος της, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και μέγα πρόβλημα ε, ξηρασίας. 10 εκατομμύρια άνθρωποι ε, πλήττονται από ε, λειψιδρία και ξηρασία στην Αιθιοπία. Αυτά για τους βραχυπρόθεσμους στόχους, για τους πιο μακροπρόθεσμους. Με χαρά να συμφωνήσω και να υπογραμμίσω και εγώ με αυτό που είπατε ότι ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε μια προοπτική ζωή για τους νέους στον τόπο τους. Ωραία όλα αυτά, αλλά γιατί δεν σας πιστεύω. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ ψηλή η ανεργία των νέων. Έχουμε δικό μας πρόγραμμα με 6 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουμε τους νέους για την εγγύηση για την νεολαία για να βρουν δουλειά και να τους βοηθήσουμε. Αλλά στην Ισπανία, στην Ελλάδα και αλλού ε, οι αριθμοί των νέων ανέργων είναι τέτοιοι ώστε εξακολουθούν να φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί για να μεταναστεύουν. Στην Ευρώπη, ε, που σε άλλες περιοχές, Βόρεια Ιταλία, Βέλγιο, ε, Ολλανδία, Γερμανία για να βρουν δουλειά γιατί στη χώρα τους δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Αν δεν καταφέρουμε να τα κάνουμε αυτά μέσα στην ίδια μας την Ευρώπη, πώς θα τα καταφέρουμε στην Αφρική. Θα τους δώσουμε και επαγγελματική, δηλαδή προοπτική. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα δημιουργήσουμε δουλειές. Εμείς δεν μπορούμε παρά να υποστηρίζουμε τις εκάστοτε κυβερνήσεις, τις προσπάθειες που κάνουν να δημιουργηθεί καλύτερο επενδυτικό κλίμα και τα λοιπά γνωστά για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Εγώ πώς το καταλαβαίνω. Πολύ αισιόδοξα μας τα λέτε. Και μήπως συγκεκριμένα παραδείγματα θα μπορούσατε να μας δώσετε για να καταλάβουμε έτσι παραδείγματα ότι καταφέραμε μαζί με τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό θα ήταν πιο πιστικό για μένα. Ευχαριστώ. Το προσφυγικό είναι κλασικό παράδειγμα αποτυχημένης αναπτυξιακής πολιτικής. Άμα είχαν αναπτυχθεί θα επικρατούσε και η ειρήνη σε αυτές τις χώρες και δεν θα υπήρχε προσφυγικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει ειρήνη, είναι ευαίσθητα αυτά τα κράτη, έχουν κατακαιρματιστεί, η διεθνή κοινότητα τίποτα δεν κάνει για να τα βοηθήσει. Έχει ως αποτέλεσμα την κατάσταση που ξέρουμε και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και είμαστε κι εμείς θύματα της αποτυχίας της διεθνούς τάξης πραγμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοένα και περισσότερα θα γίνει ο στόχος αυτών των ανθρώπων που είναι ξαναλέω απόρριοι αυτής της αποτυχίας. Και εγώ την αποδίδω αυτή την αποτυχία πλήρως στα Ηνωμένα Έθνη. Τίποτα δεν έκαναν, απολύτως τίποτα, τα τελευταία πέντε με 6 χρόνια. Ξέρω ότι δεν είναι ε, σωστή στιγμή τώρα, ε, γιατί έχει δεχθεί τόσες επικρίσεις ε, ο ύπατος εκπρόσωπος και είπαμε ότι ε, είπαμε επίση ότι θα έπρεπε, είναι και ευθύνη των ε, χώριων ε, κυβερνήσεων. Πρέπει εκεί να προστατεύσουν του επικόστου. Υπάρχει αυτή η αντίληψη στη διεθνή πολιτική για την ανθρωπιστική δράση, αλλά τελικά τα πετάξαμε πλέον τώρα όλα στη θάλασσα. Δηλαδή τι λέμε, αφήστε του. Στην τύχη τους να πάνε να πνιγούν και εμεί να κοιτάξουμε τώρα τι μα συμβαίνει γιατί έχουμε εκατομμύρια πρόσφυγε που έρχονται σε εμά. ή θα αναθεωρήσουμε πλήρως αυτά, αυτές τις παρεμβάσεις μας ε, και θα αναθεωρήσουμε την άποψή μας σε σχέση με την ευθύνη που έχουμε να τις προστατεύσουμε ή να χτίσουμε ένα πελώριο τείχο και δεν θα μας νοιάζει τι γίνεται πέρα από αυτό. There ε, ε, από την ε, εμπειρία μας βλέπουμε ότι αυτό, αυτή την επιλογή την έχουν κάνει πολλές χώρες. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Έχουμε όμως επιλογή και αυτό μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να εξακολουθήσουμε να κάνουμε είναι να δεχθούμε τις επιπτώσεις αυτής της αποτυχημένης, αποτυχημένης πολιτικής, αλλονών η αποτυχία, δεν είναι δική μας, και να πληρώσουν πάλι φορολογούμενοι. Παράδειγμα. Μήπω αυτά που γίνονται τώρα στη Συρία θα, θα συμβούν και στην Αίγυπτο. Μπορεί κάποιο να το διανοηθεί αυτό. 20 εκατομμύρια πρόσφυγες θα έχουμε άμα συμβεί κάτι τέτοιο. Και κάνουμε εμεί τίποτα αυτή τη στιγμή για να το αποτρέψουμε. Ή να κατανοήσουμε τουλάχιστον τι επιπτώσει ενός τέτοιου φαινομένου αν προκύψει. Όχι, περιμένουμε απλώ. Τίποτα, άπραγοι, περιμένουμε. Τι θα κάνουμε άμα ε, μας φορτώσουν 20 εκατομμύρια Αιγύπτους ε, στην Ευρώπη. Τι θα κάνουμε τότε. Now, the next big issue. Το άλλο μείζον θέμα είναι η Αφρική. Αναπτύσσεται η Αφρική και θα γίνει οικονομικός γίγαντας. Όμως υπάρχουν και αποτυχημένα κράτη στην Αφρική ταυτόχρονα και Έχουμε τη σύμβαση ΛΟΜΕ τη χώρες εκεί 25 χρόνια τα ίδια κάνουμε εκεί πέρα και παρότι έχουμε αυτούς τους εταίρους και προσπαθούμε να επιτύχουμε ευημερία σε εκείνους, ούτως ώστε, ε, επιτόπου, ούτως ώστε να μην έρθουν στη γυραιά Ήπειρο. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό στο μέλλον. Και γι' αυτό Τώρα λέω τα δικά μου βέβαια. Ε, ο Στεφάνο, εγώ ε, και οι άλλοι είχαμε τη φαϊνή ιδέα ε, να απελευθερώσουμε τα ταμεία τα αναπτυξιακά, ούτω ώστε Έχουμε τα 60 δις, έτσι, στην πρώτη φάση και μετά 200-300 ίσως δις για, στη συνέχεια μεταγενέστερα για να επενδύσουμε στην Αφρική και αλλού ούτω ώστε πραγματικά να δημιουργήσουμε επιχειρηματικό κλίμα, θέσεις εργασίας κτλ. Για να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας. Βαρέθηκα πια. Γιατί κανείς εδώ στο κοινοβούλιο δεν κατάλαβε ποτέ ότι ο στόχος που επιδιώκουμε είναι win-win, ε, ε, αμοιβαίω επωφελής. Δεν είναι ότι τα παίρνουμε από τους δικούς μας και τα δίνουμε στους στοχούς. Ε, αυτό το μήνυμα θέλ, θέλουν κάποιοι ε, να περάσουν. Όχι. Είναι επωφελές και για μα. διότι δημιουργούμε ευκαιρίες σε αυτές τις χώρες και κερδίζουμε από αυτό. Σε αυτή την Επιτροπή όμω ποτέ δεν επικράτησε αυτή η άποψη και ως αποτέλεσμα στην Επιτροπή Εμπορίου ε, ένα ολόκληρο συνάφι και τροφοδοτεί τον αναπτυξιακό μηχανισμό που επιταχύνει την ανάπτυξη παρότι τι να πω που δεκάρα τίποτα δεν, δεν ασχολούνται καν με τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουμε θέσει εμείς. Όσο λοιπόν σου επιτρέπουμε να προωθούν μόνο εμπορικούς στόχους, δηλαδή άλλη επιτροπή, ενώ είναι ο πρώτος, η κινητήριος δύναμη για να επιτύχουμε ανάπτυξη, άλλοι αποφασίζουν. Όσο λοιπόν το επιτρέπουν να συμβαίνει αυτό, θα έχουμε σοβαρότατα προβλήματα. Έχουμε, μελέτη δεν χρειαζόμαστε, ξέρουμε τι δεν πάει καλά, τι θα κάνουμε είναι το θέμα. Να πάει διάσκεψη των πρόεδρων ή πρόεδρος μας και να τους πει ότι τώρα που έχει φτάσει ε, σε αυτό το σημείο η κατάσταση, εμείς θα επιφορτιστούμε με τα ζητήματα τα εμπορικά. Τα εμπορικά που χρησιμοποιούμε για να υλοποιήσουμε αναπτυξιακή πολιτική. Δεν μπορούμε να έχουμε εμεί σχέσει με τι αναπτυσσόμενε χώρε και αφήνουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε ε, στι εμπορικέ του σχέσει να πηγαίνουν στην άλλη επιτροπή. Μόνο τότε θα συνδυάσουμε τα αναπτυξιακά μα προγράμματα, γιατί προσπαθούμε να διοικητεύσουμε τα κονδύλια, χωρί όμω τι εμπορικέ πολιτικέ. Δεν γίνεται αυτό, διότι πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο με ολιστικό τρόπο. Αλλιώ, ε, όπω και όλα τα υπόλοιπα, θα είναι κατακαιρματισμένη η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, Νίρ. Αυτό είναι το θέμα για τη σύσταση των νέων επιτρόπων ε, Χόλμπρου και Αλλιώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Καταρχήν, η αναπτυξιακή πολιτική ε, προσανατολίζεται στην καταπολέμηση της φτώχειας και όχι, πώς να το πω τώρα, τη διεθνή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Και τώρα, αν μας απασχολεί η καταπολέμηση των αιτίων ε, της ε, φυγής, αυτό είναι μακράς πνοής. Μιλήσατε κι εσείς για την καταπολέμηση της ανεργίας, ε, να δούμε και άλλες αιτίες, συστημική σύνδεση τους και εξάρτηση. Τώρα όμως αν βγαίνουμε και φτιάχνουμε διάφορα ταμεία, καταπιστεύματα, παίρνουμε από εδώ λεφτά, κάνουμε μεταφορές πιστώσεων, τα λεγόμενα ευέλικτα κιόλας μέσα έχουμε μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά ως προς τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Και έχει νόημα όταν τα προγράμματα αλλά και τα θέματα είναι τόσο μακροπρόθεσμα να είναι τέτοια τακτική μας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η άμεση ερεσιμότητα που έχει ξεπεραστεί και στην πράξη και στη λογική. Υπάρχουν και κάποιες αρχές ε, αποτελεσματικότητα αναπτυξιακή βοήθεια, βοήθειας, ε, η έννοια του ownership, δηλαδή να το ε, στενίζονται και να το κάνουν κτήμα τους αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Και τι γίνεται με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εμείς πώς ελέγχουμε αυτά τα χρήματα. Βγαίνουμε και κάνουμε διάφορες συμφωνίες, deal κανονικά με την Τουρκία τώρα, που είναι εκτό τη συνήθους κοινοβουλευτική και δημοσιονομική διαδικασία. Άρα εκφεύγει αυτό και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τέτοια πράγματα δεν είναι σωστά. Μπορεί να χρειάζονται τέτοιε συμφωνίε σε έκτακτες περιστάσεις, αλλά ε, εσεί είπατε ότι η συμπεριφορά μας τώρα δεν ε, υπαγορεύεται από ε, την έκτακτη και επίγουσα ανάγκη, αλλά ε, επιταχύνεται. Αν είναι αυτό να γίνει κανονικότητα όμως, χρειάζονται συνήθεις διαδικασίες για τον προπολογισμό και να μπορεί και το Κοινοβούλιο να ασκεί τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο. Το είπε και ο Νόρμπερτ Νόιζερ. Ε, δεν είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ αφηρημένα είναι αυτά που μας λέτε και τελικά δεν ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά. Και ένα τελευταίο. Τώρα η προσέγγιση μας βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην πολιτική μετανάστευση. Αλλά συνολικά στις σχέσεις μας με τις ίδιες χώρες ισχύει το ίδιο. Τώρα, όταν μιλάμε για απέλαση ή επαναπροωθήση, μιλήσατε για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ε, μένουν παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να απελάβνονται. Αν γίνεται αυτό πάρα πολύ γρήγορα, πώς θα συμβεί. Και γνώμονα δεν είναι πάντα η ασφάλεια, ούτε η αξιοπρέπεια, γιατί μιλάμε για συνέχεια για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών, ούτε είναι δεδομένη. Και κατά πόσο είναι ασφαλείς και ζουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι σε τέτοιες χώρες, σε αυτές που τους επαναπροωθούμε. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Χρειάζονται νόμιμες οδοί και ασφαλείς οδοί ε, ε, διαφυγής. Ε, είναι πάρα πολύ λίγες αυτές οι νόμιμες και κάτι πρέπει να κάνουμε και μάλιστα πολλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλιό. Euh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Πολλά πράγματα θα μπορούσα να πω επί της ουσίας όπως και ο κύριος Δέβα, έτσι και εγώ, νομίζω ότι συστηματικά ασχολούμαστε μόνο με τις συνέπειες και όχι με τα αίτια, τα βαθύτερα αίτια της κατάστασης αυτής που έχουμε σήμερα στον πλανήτη. Έχουμε όλα αυτά τα νέα μέσα, όλα αυτά τα ταμεία, λοιπόν, ποιας πολιτικής τελικά. Αν τελικά ο απότερος στόχος είναι να καταλήγουμε στην κατάσταση αυτή που έχουμε στη Μέση Ανατολή, στη φτώχεια αυτή που έχουμε στην Αφρική. Για πόσα χρόνια θα δίνουμε ακόμα χρήματα στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας που δεν βοηθούν τελικά τους φτωχούς αυτούς πληθυσμούς να απτυχθούν 40 ολόκληρα χρόνια. Δίνουμε κονδύλια σε ηγέτες οι οποίοι βρίσκονται ακόμα στη θέση τους μετά από όλα αυτά τα χρόνια και για παράδειγμα στην έκθεση αυτή θα μπορούσαμε να μιλούσαμε περισσότερο για πολιτικό πλουραλισμό ή ακόμα και για δημοκρατική εναλλαγή ή ακόμα απλώς και για εναλλαγή όσον αφορά την εξουσία. Και αν δούμε πώς έχουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Για το Κονκό Μπραζαβίλη τέθη το ζήτημα πριν από λίγες ημέρες και νομίζω ότι είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή ότι εξακολουθούμε και έχουμε τον ίδιο ηγέτη, μόλον ότι υπήρχε τέτοια τεράστια αναταραχή γύρω από τις εκλογές και συνεχίζεται παράλληλα η ενδειξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είχε συμβεί τίποτα, ενώ παράλληλα δεν έχουμε υποδομές στη χώρα αυτή, δεν υπάρχουν σχολεία, μειώνεται ο αριθμός των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο, έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα βίας κτλ. Και έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι από τη χώρα αυτή και από άλλες χώρες προκειμένου να λάβουν υγειονομική υπερίθαλψη εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα έπρεπε στη χώρα τους να έχουν τις απαραίτητες υποδομές. Όσον αφορά τώρα την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας θα έπρεπε να ήταν μια πολιτική η οποία θα εξισορροπούσε τις μετακινήσεις στον πλανήτη. Πάντα θα έχουμε τέτοιες ροές. Και πάλι όμως δεν θα έπρεπε εμείς να συμβάλλουμε, αν θέλετε, στην έλλειψη τάξης, στη Λιβύα, η Γαλλία, και μιλώ βέβαια εξ ονόματος της χώρας αυτής που εκπροσωπώ, φέρει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Κανείς δεν τολμά να το πει αυτό. Αν δεν είχαν επέμβει στην Λιβύη, δεν θα είχαμε τότε την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα. Πλήρης αναρχία. Και λέμε ναι, θα έπρεπε να έχει σταματήσει, έπρεπε να βγάλουμε από τη μέση τον Καντάφη. Ναι, ωραία. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε παράλληλα να έπρεπε να σεβαστεί περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και σε πολλέ άλλε χώρε, όπω για παράδειγμα στην Κίνα. Τίθεται λοιπόν σαφώ το δημοκρατικό ζήτημα, καθώ επίση και το ζήτημα των αξιών που θα πρέπει να διέπουν την απτυξιακή μας βοήθεια. Μένα μου φαίνεται λογικό να έχουμε προϋποθέσεις προκειμένου να δώσουμε τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου προς τρίτες χώρες, ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους στόχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό το πράγμα, διαφορετικά τα χρήματα αυτά δεν θα πιάσουν πουθενά τόπο, θα καταλήξουν μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ηγετών των, των ηγετών των χωρών αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι η αιρεσιμότητα είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Ερεσιμότητα που θα πρέπει να συνδέεται με τη χρηστή μη διακυβέρνηση των ανθρώπων αυτών απέναντι στις χώρες τους και στον πληθυσμό τους. Και κάτι ακόμα για ποιο λόγο θα πρέπει να συμβάλλει συνεχώς ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, για ποιο λόγο να μην μιλήσουμε και για τις μεγάλες βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμα και τις μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες και τις μεγάλες δημόσιες βιομηχανίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα, ή της ενέργειας. Δεν θα μπορούσαν και αυτές με τη σειρά τους να συμβάλλουν. Νομίζω ότι και αυτό αποτελεί μέρος της ανισότητας και της αδικίας που όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες καταδεικνύουν αυτή τη στιγμή, τονίζουν αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σημαντικό να μας απασχολήσουν τα ζητήματα αυτά, γιατί όσο δεν τα θεραπεύουμε, όλο και θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Και όπως είπε ο κύριος Σεντέβα, δεν είναι μόνο η Αίγυπτος, αλλά και σε άλλε χώρε του Μαγκρέπ, για παράδειγμα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ανάλογα προβλήματα. Αν έχουμε τέτοια πολιτικά προβλήματα στι χώρε αυτέ, τι θα κάνουμε με τα εκατομμύρια μεταναστών που θα φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα θα σταματήσει πλέον να είναι μόνο ευρωπαϊκό, θα είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ένα παγκόσμιο πρόβλημα φτώχεια, εξαθλίωση που θα οδηγήσει σε πολέμου. Προφανώ δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιμέρους κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθούν συγκεκριμένα όρια, περιορισμούς και προϋποθέσεις για την αντιξιακή πολιτική. Γιατί αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε θα επιστρέφουμε συνεχώς κάθε χρόνο στην Επιτροπή αυτή συζητώντας τα ίδια προβλήματα χωρίς να καταφέρνουμε να βρούμε καμία απολύτως λύση. Ευχαριστώ. Τώρα ακολουθούν μιλητές οι υπόλοιποι. Είχαμε έναν από κάθε πολιτική ομάδα, οι υπόλοιποι δίλεπτο. Ε, η κυρία Σλάιν, η Χάουταλα, ο κύριος Φροντσουλίκα, η Γιώδης Αρσεντίνη και η Πατρίσια Τόγια. Um, Ευχαριστώ. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε δει, μας δόθηκε ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα και όπως είπα και τότε, Φυσικά χρειαζόμαστε ένα, ένα επενδυτικό πρόγραμμα ε, στην Αφρική και φυσικά χρειαζόμαστε ανανοημένε εταιρικέ σχέσει με αφρικανικέ χώρε. Διαβάζοντα όμω αυτή την ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Είχα την ευκαιρία ότι ασχολούμαστε με τη φύλαξη των συνόρων, την ανάπτυξη ενδογενών ικανοτήτων και φυσικά τι επιστροφέ. Ε, η αιρεσιμότητα είναι ξεκάθαρη και για τα σύμφωνα αυτά θα φροντίσει λίγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων σε όλα τα κομβικά σημεία να υπάρχουν ε, θετικέ επιπτώσει επί των μεταναστευτικών ροών και θα μεγιστοποιήσει τι προσπάθειε στο θέμα διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ξέρετε, ο, όπως είπαν και οι συναδελφοί, ότι στο άρθρο 209 της Συνθήκης Λισαβόνας ξεκάθαρα υπάρχει αναφορά σε αυτό. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο, στη συνεργασία που έχει την αναπτυξιακή πολιτική πρωταρχικό στόχο έχει τη μείωση και μακροπρόθεσμα την εκρίζωση της φτώχειας και επίσης ε, την ε, ουδετερότητα ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό όμως διακυβεύεται εδώ και φοβάμαι ότι άμα ε, πανιεραρχηθούν οι προτεραιότητες μας στην αναπτυξιακή πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση θα θέσει εν κινδύνο τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουμε για την εκρίζωση της φτώχειας των ανισοτήτων και των βασικών αιτιών όπως τα λέτε και εσείς root causes στα αγγλικά της μετανάστευσης. Η διαφύλαξη των, η φύλαξη των συνόρων δεν εξυπηρετεί αυτούς τους στόχους. Δεν έχει σχέση με τη φτώχεια και τις ανισότητες. Και ξαναλέω, ο πρωταρχικός στόχος, όπως διαγράφεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μεν η διάσωση των ζώων, όμως δυστυχώς δεν είναι η σε με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αυτές τις εταιρικές σχέσεις. Άλλα είπε το Συμβούλιο πριν από δύο εβδομάδες, γιατί ο, ο πρωταρχικός στόχος, τι λέει το Συμβούλιο, διαβάζω, είναι οι επιστροφές πρωταρχικός στόχος, προτεραιότητα, ύψιστη προτεραιότητα. Δεν βλέπω στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τίποτα για διασώσεις ε, και δεν βλέπω τη σχέση με τη δική σας ανακοίνωση για τα κονδύλια. Έχουμε επιπλέον ε, ε, δεσμεύσεις, ε, ανάληψη υποχρεώσεων και αν κατάλαβα καλά, άλλα 500 εκατομμύρια θα μπουν στο καταπίστευμα, τα πάρουμε από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και 3,1 δις είναι η προποδότηση, θα, θα τα πάρουμε από, το, από την Facility, το χρηματοδοτικό μέσα για την πολιτική γειτονία από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Ναι, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, δεν δηλαδή, τι κάνουμε. έχουμε την εκτροπή κεφαλαίων που ε, κανονικά θα θυγετεύονταν στους πλέον αδυνάμους. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ο καλύτερος τρόπος και για τις νόμους οδούς μεταναστευσής. Δεν ξέρω, για τα... υπάρχει ένα μόνο μέσο για να μην πέσουν στα χέρια των διακινητών ε, οι άνθρωποι, το είπε και η Μογκερίνη, να δημιουργηθούν περισσότερες, ε, περισσότεροι νόμιμοι τρόποι μετανάστευσης και ταυτόχρονα κατοχυρωθεί ο έλεγχος, ο μέγιστος δυνατός έλεγχος από το Κοινοβούλιο. Γιατί αλλιώ δεν βλέπω να έχετε υποστήριξη για τα σχέδιά σα. Ευχαριστούμε, Χέντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό. Να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μεγάλο σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή μας πολιτική. Με κάθε σεβασμό για τα λεγόμενά σας, κύριε Γενική Διευθυντά, μιλήσατε για στόχους που έχουν να κάνουν κατά κλιματικής αλλαγής, κατά πολέμηση ενεργείας των νέων, παιδεία, εκπαίδευση. Αυτά που προτείνεται να γίνουν με διάφορους τρόπους, είτε στον προϋπολογισμό, είτε με τροπολογίες, ε, contributing to peace and ε, για την σταθερότητα, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι απεμπολούμε τις αρχές ε, της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες. Προχωρούμε σε κινδυνολογία, σε κοντόφθαλμες λύσεις, βραχυπρόθεσμες κτλ. σε σχέση με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Ας μην μιλάμε λοιπόν για μακροπρόθεσμα αν ε, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση μόνο με βραχυπρόθεσμα μέτρα. Με πολύ μεγάλη θλίψη το λέω αυτό. Έχω την αίσθηση ότι η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απαχθεί και είναι όμοιρος, όχι στο βωμό ε, άλλων πολιτικών. Δηλαδή δεν αλλάζουμε τις πολιτικές της γεωργίας ή ε, άλλου είδους του εμπορίου για να μπορεί ο κόσμος να μένει στον τόπο του, αλλά ε, μια ομοιρία στο βωμό ε, ε, ενός θέματος που είναι άσχετο και ξένο προς την απτυξιακή βοήθεια. Μιλάτε για την καταπολέμηση της νέας μετανάστευσης, ε, να προωθήσετε, λέτε, νόμιμες οδούς, αλλά μακροπρόθεσμα θέλετε να το κόψετε και αυτό. Λέτε ότι θα βοηθάμε τις χώρες να αυτοβοηθούνται, ξέρω εγώ, Συναχινά και Χειρακίνη, αλλά όλο και περισσότερο βάζετε στην αναπτυξιακή βοήθεια όρους για να έχετε περισσότερους ελέγχους που είναι πάρα πολύ ξένο προς την αρχή ε, του σεβασμού των εταίρων της αναπτυξιακής βοήθειας. Και επίσης, δεν πιστεύω, αγαπητέ κύριε Ντέβα, ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενδιαφέρεται για μας το Aid for Trade, για εμπόριο αναπτυξιακή βοήθεια για την πρόθεση του εμπορίου. Δεν με πειράζει αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να κυριαρχήσει το εμπόριο και να καταστραφεί η αναπτυξιακή βοήθεια. Και πού πηγαίνουμε και το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Και τα χρήματα πού πάνε. Σε αλότριους ε, σκοπούς που δεν έχουν και σχέση, ούτε συμμορφούνται με τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως εξήγησε η Έλλη Σλάιν, δεν σας κρύβω την ανησυχία μου. Χρειαζόμαστε μια συζήτηση επί τη αρχή για το τι συμβαίνει πραγματικά για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Με αυτές τις ε, κατακαιρματισμένε και αποσπασματικέ αλλαγέ νομίζω έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Ο κύριος Φροντσούλικα. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Ανέκαθεν πίστευα ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι μία από τις σημαντικότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε μία φυσιολογική ζωή που θα έπρεπε να ζει ένας άνθρωπος όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. Όπως υπόθηκε πριν από λίγο, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέα οχυρά με υψηλούς στίχους και να απομονωθούμε από όλους τους υπόλοιπου. Τα προγράμματα ανάπτυξης για όλες τις χώρες αυτές είχαν ως απότερο στόχο να βοηθήσουν τις χώρες αυτές να αναπτυχθούν πραγματικά, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, αλλά τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να επιβάλλει τίποτα το θετικό στις χώρες αυτές που λάβανε δισεκατομμύρια ευρώ. Κατα... Αποτύχαμε να επιβάλλουμε το κράτος δικαίου, την πραγματική δημοκρατία, τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω, ούτως καθεξής αποτύχαμε σε όλα αυτά. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ξέσπασε η κρίση η μεταναστευτική, η οποία επηρεάζει τα πάντα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα έχετε συνειδητοποιήσει τι συνέβη με τον Brexit, όπου πολλοί Βρετανοί πολίτες ψήφισαν υπέρ του Brexit εξαιτία τη μετανάστευσης, εξαιτία της τρομοκρατίας που συνδέεται με τη μετανάστευση και το καθεξής. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα όλα αυτά τα ζητήματα βρίσκεται σε πολύ δεινή θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλήττεται από πάρα πολλές συγκρούσεις γύρω της. Πρέπει λοιπόν να καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ένα τον άλλο τρόπο να επιλύσει τα προβλήματα που βλέπει αυτή τη στιγμή τόσο στη Μεσόγειο και στην Ανατολικά της και να βοηθήσει έπειτα στην ανοικοδόμηση αυτών των περιοχών. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, εκατοντάδες εκατομμύρια νέοι στην Αφρική, στη Μέση στην Ανατολή δεν έχουν θέση απασχόλησης. Και τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Κοιτάνε προς την Ευρώπη. Επιθυμούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το φαινόμενο αυτό ακόμα εμείς δεν έχουμε όμως κάποια στρατηγική. Συζητήσαμε την υπόσχεση του κύριου Γιούνκερ 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στη συνδιάσκεψη της Μάλτας για την αντιμετώπιση της προσφαιρικής κρίσης και στη συνέχεια αρχίσαμε να παραπονιόμαστε γιατί αυξήθηκε το ποσό εκείνο το οποίο θα έπρεπε να δοθεί προς την Τουρκία. Εκφτάσαμε ακόμα και τα 6 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε λοιπόν να λογοδοτήσουμε για τα χρήματα αυτά απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας ζητούν να δουν πώς θα καταφέρουμε εμείς να, να αντιμετωπίσουμε την μεταναστευτική αυτή κρίση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε χώρο όπως η Τινησία, το Μαλί, ο Νίγηρα, η Νιγηρία ή ακόμα και η Ερυθρέα, η Αιθιοπία. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε αποτύχει. Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική προκειμένου να έχουμε μια βαθύτερη ολοκλήρωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι σήκωναν πλακάτ σε κάποιε διαδηλώσει πρόσφατα λέγοντα η Ευρωπαϊκή Ένωση για του Ευρωπαίου μόνο. Και αυτό πρέπει να το αφουγκραστούμε σαν μήνυμα. Παράλληλα, χρειαζόμαστε όμω μία στρατηγική προκειμένου να ισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ ημών και να έχουμε και μία κοινή στρατηγική απέναντι στη μετανάστευση, η οποία δυστυχώ δεν υπάρχει ακόμα. Σα ευχαριστούμε πολύ. κυρία Σαρτζετίνη έχει το λόγο και μετά η κυρία Τόια πρώτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Μανσερβίση, σα άκουσα και προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό για το, ρόλο του ελέγχου ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και τα λοιπά από την Επιτροπή μας. Είδαμε όλα τα στατηγικά έγγραφα στις χώρες, για τις χώρες ΑΚΕ τα τελευταία χρόνια και τα ελέγχαμε. Και τώρα υπάρχουν προτάσεις στην ανακοίνωσή σας θολές και ασαφείς ως προς το τι γίνεται. Και λέτε να επαναδρομολογηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό, το Κοινοβούλιο πότε θα δει αυτέ προτάσει για να μπορεί ξανά να ελέγχει το Ταμείο. Γιατί το λέω αυτό, διότι στι προηγούμενε συμφωνίε, τα deal τύπου Τουρκία, έχει συναυθεί με τέτοιο τρόπο η συμφωνία που δεν χωράει πουθενά κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οπότε, παρακαλώ να το διευκρινίσετε αυτό. Επίση, υπό το φως των διεθνών δεσμεύσεων για ε, την ανάπτυξη. Το 7 το 0,7% ξέρετε του ΟΑΕΠ ε, που προβλεπόταν, ποια, ε, ποιο κράτος μέλος θα τηρεί αυτό. Αυτή τη συζήτηση κάνουμε χρόνια ολόκληρα. βλέπουμε να μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση και επίσης βλέπουμε στην πρόταση που μας κάνετε τώρα ερεσιμότητα να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό ότι δεν θα πρέπει βοήθεια να συνδέεται με όρους και προϋποθέσεις. Καμία σχέση δεν έχει με την καταπολέμηση και την εκρίζωση της φτώχειας αυτό. Η παρούσα πρόταση, η ανακοίνωση και πάλι συνδέει την ε, ε, βοήθεια ε, με αυτό. Εσείς έχετε περάσει από πολλά πόστα. Σα θυμάμαι στην Γενική Διεύθυνση Ιστορικών. Τώρα έχετε αλλάξει η Γενική Διεύθυνση, έχετε φύγει από εκεί. Υποτίθεται ότι προστατεύετε την αναπτυξιακή βοήθεια για να πηγαίνει εκεί που έχει ε, προβλεφθεί άρθρα 21 και άρθρα 208. Οι κείμενες ε, προτάσεις δεν σέβονται τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και μια τελευταία παρατήρηση, για τις επιστροφές. Δεν υπάρχουν προτάσεις στην ανακοίνωση για επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής που δεν είναι και δικό μας θέμα, είναι της ΛΥΜΠΕ. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν προτάσεις. Άρα, εγώ πώς το κατανοώ. Προσπαθούμε να οργανώσουμε τις επιστροφές μέσω ε, χρηματοδοτικών κινήτρων από το ODA. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτά. Από ODA που είναι επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια κρατική. Σταματήστε λοιπόν να συζητάτε την ιδεολογία και κάντε αυτό που χρειάζεται, κοινοβουλευτικό έλεγχο που δεν γίνεται τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Η Πατρίσια Τόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι η δική μου προσέγγιση είναι διαφορετική από τους υπόλοιπους συναδέλφους που άκουσα εδώ πέρα σήμερα στην Επιτροπή μας. Εγώ εξετάζοντας την ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σαφώς έχει ένα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, ακόμα και διόρθωση σε κάποια σημεία, θεώρησα ότι θα πρέπει να διατηρήσω μια θετική στάση. Συντοποιούμε όλοι, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ζούμε, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω μας και το πώς είναι επίγους ανάγκη να καταφέρουμε να συνδυάσουμε ανάπτυξη και εξωτερική πολιτική προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε γύρω μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε όχι τόσο τις νομικές πτυχές, αλλά τα ουσιαστικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια τη δημοκρατία, το καθεστώς δημοκρατίας σε κάποιες χώρες. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά, τότε πραγματικά θα πληγεί ακόμα και η ίδια η δημοκρατία και οι κοινωνικές συνθήκες στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μου κάνει εντύπωση που δεν καταφέρατε να το δείτε αυτό περισσότερο στα πλαίσια της ανακοίνωσης αυτής, που δικαιολογούν τελικά και τους ίδιους τους στόχους της ανακοίνωσης αυτής όπου έχουμε, αν θέλετε, και τις βασικές μας αρχές στα πλαίσια της συνεργασίας. Μέχρι στιγμής, η πολιτική αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωση όντω δεν είχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Δεν είχαμε θέσει του σωστού στόχους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να επαναπροσανατολίσουμε την πολιτική αυτή. Να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια νέα τέτοια πολιτική, να έχουμε μια αναπτυξιακή συνεργασία η οποία θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα, που θα μπορούσε όντω να συμβάλλει στη μείωση τη φτώχεια, στη μείωση τη ένδυα ή να συμβάλλει και στα δημοκρατικά πολιτεύματα. Δεν το έχουμε πετύχει όμω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κατάσταση με καινοτόμε λύσει. Να δούμε για παράδειγμα τα, βαθύτερα αίτια. Όντω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε για όλες τις πολιτικές να δούμε ποια είναι τα βαθύτερα αίτια, όχι μόνο για τη μετανάστευση, αλλά να καταφέρουμε να επαναπροσανατολίσουμε πιο αποτελεσματικά και την ίδια την εμπρεξιακή πολιτική. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε, να αποσαφηνίσουμε κάποια σημεία. Θα αναφερθώ σε ένα εγώ, το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Να δούμε τι θα γίνει με τους σπόρους οι πόροι οι οποίοι δεν είναι αρκετοί και προσπαθούμε να βρούμε δημιουργώντας νέα χρηματοδοτικά μέσα. Πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στο σημείο αυτό. Ξέρετε ότι όταν μιλάμε για το επενδυτικό πρόγραμμα Juncker για όλα τα νέα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτημα αυτό μας απασχολεί. Πρέπει να μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο τώρα. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο ενδελεχής έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς θα γίνει όμως κάτι τέτοιο, πώς θα καταφέρουμε να συντονίσουμε τελικά όλα αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα. Πώς θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια νέα χρηματοδοτική πολιτική για την αναπτυξιακή συνεργασία. Πώ θα καταφέρουμε να έχουμε περισσότερη σαφήνεια στα νέα αυτά μέσα. Ευχαριστώ. Κύριε Τσέλλερ, τελευταία στιγμή ήρθατε δίλεπτο το πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η συζήτηση τώρα έχει μπει στι τροχέ που κανονικά θα έπρεπε να ήταν. Πόσο αποτελεσματική δηλαδή ήταν η αναπτυξιακή μα βοήθεια τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε. Και τι γίνεται με τα σημερινά γεγονότα. Θέλω και εγώ να σας προειδοποιήσω για τις ψευδεστήσεις. Στη Γερμανία ακούμε τώρα στοιχεία που λένε ότι τους τελευταίους 14 μήνες δεχτήκαμε πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και σε μια αγορά εργασία που πάνω κάτω λειτουργεί καλά ε, απορροφήθηκαν 30.000 από το 1 εκατομμύριο. 30.000 βρήκανε δουλειά από 1 εκατομμύριο. Ε, καταλαβαίνετε. Είναι αυτό νόητα τα στοιχεία και μιλούν από μόνα τους. Έχω άλλη ερώτηση όμως για την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποκρινόμαστε ότι ε, μπορούμε να επηρεάσουμε πολλές από τις χώρες αυτές που τις ε, κατατάσσουμε στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων ακόμα κρατών και βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αυξήσει τη μακροοικονομική βοήθεια προς τα κράτη αυτά. Αυτό έχει νόημα μόνο εφόσον ταυτόχρονα ε, λαμβάνετε μέρημνα ή το έχετε συμφωνήσει με τις χώρες αυτές να ενισχύσουν τη δική τους ε, δημοσιονομική βάση και να την βελτιώνουν. Αν προσπαθούμε εμείς όμως νομισματικά συστήματα ε, σε τέτοιες χώρες να τις υποστηρίζουμε με μακροοικονομική βοήθεια, αλλά τα κέρδη να εξακολουθούν να τα μεταφέρουν σε ε, διεθνείς ε, οάσεις, ε, φορολογικούς παραδείσους και τέτοιες τράπεζες, δηλαδή φεύγουν από τη χώρα τα κέρδη αυτά, τότε τι να την κάνουν τη μακροοικονομική βοήθεια, δεν έχει νόημα. Διαβάζω ότι η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό σκέφτεται αυτό τον καιρό να επιβάλλει στις διεθνείς εξορρεκτικές εταιρείες ε, μια ρύθμιση, μάλλον να τους επιτύψει το ΦΠΑ, γιατί τους λένε ότι θα σηκωθούν να φύγουν αν ε, τους επιβάλλουμε ΦΠΑ. Οπότε, έτσι κι αλλιώς, τη λαιλατούν που τη λαιλατούν τη χώρα, ε, θα τους κόβουν και θα τους χαρίζουν το ΦΠΑ τώρα. Πώς θα μπορέσει να ορθοποδήσει μια τέτοια χώρα. Αυτό θέλουμε. Έχετε σκεφτεί τι κάνουμε όταν δίνουμε μακροοικονομική βοήθεια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουμε εμείς τι τα κάνουν αυτά τα λεφτά στις χώρες. Δεν θα πρέπει να καταβάλουν και εκείνοι προσπάθειες έτσι ώστε να βάλουν σε μια τάξη τα δημόσια οικονομικά τους και τα φορολογικά τους έσοδα. Κατά τα άλλα είναι μια τρύπα στο νερό όλα αυτά. Thank you. I just have... Ευχαριστώ. Ε, να πω και εγώ δύο πράγματα. Πότε μπορούμε να περιμένουμε το, την πρώτη τέτοια συμφωνία ε, compact. Ε, προσπαθώ να καταλάβω πώς θα είναι. Θα, πάρουμε νέα λεφτά, θα, δηλαδή θα, θα φέρνουν νέα κονδύλια και συν, ε, επιπροσθέτως θα έρθει αυτή η συμφωνία ή θα ενσωματωθούν αυτά τα επιπρόσθετα κονδύλια μέσα στο μνημόνιο, μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Ε, τώρα πέρα από το εξωτερικό επενδυτικό μας πρόγραμμα, γιατί μιλάμε για 62 δις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τρία δις που μας λείπουν από τράσφαν για την Αφρική. Μήπως θα ήταν καλύτερα να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους, οποίους και θα υλοποιούμε και μόλις ε, τα υλοποιήσουμε και μετά να περάσουμε στα επόμενα, όχι να έχουμε αυτούς τους μεγαλεπίβολους στόχους, γιατί έτσι ε, πάντοτε δίνουμε την εντύπωση ότι ε, ε, είμαστε μεγαλόστομοι, αλλά τελικά στην, ε, ε δεν ε, επιτυχάνουμε αυτές τις αλλαγές ε, που υποσχόμαστε. Απάντης. Ευχαριστώ για τα επικοδομητικά, επικριτικά σας σχόλια. Είναι πολύ χρήσιμα, είναι μέρος της ε, διαδικασίας. Να αρχίσω με αυτό που μας είπε η κυρία Σατζεντίνη. Ήμουνα στη ΔΕΛΤΑ αλλά πριν ήμουνα στην ΤΕΦΚ. Ε, ε, ασχολήθηκα χρόνια με την αναπτυξιακή πολιτική. Και αυτά που εγώ έμαθα στην προηγούμενη ζωή μου, στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ανάπτυξης, γιατί το βλέπω το, ε, το πρόβλημα από, και από τις δύο πλευρές των συνόρων, καταλαβαίνετε. Δεν είπα ότι χρησιμοποιώ μόνο την εμπειρία μου στην DG Home για να λύσω το πρόβλημα στην Αφρική. Λέω απλώς ότι είναι περίπλοκο και πολυδιάστατο το ζήτημα. Και προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου. Αν υπάρξει υποψία ότι ξαφνικά, ή μάλλον όχι ξαφνικά, αλλά έχουμε μια real politik και πλέον και ότι πάμε να κλείσουμε όλους τους δρόμους, όλους τους οδούς μετανάστευσης και προσπαθούμε προσπαθούμε, λένε κάποιοι, να φτιάξουμε φράχτες, ε, τι ήχους ε, για να τους αποτρέψουμε τους ανθρώπους. Και αν πιστέψει κάποιος ότι αυτή είναι η λύση που προτείνουμε, νομίζω ότι κάνει λάθος, διότι δεν είπαμε αυτό στην ανακοίνωσή μας. Διότι μιλήσαμε για συνένεση στην Ευρωπαϊκή Συνολική Στρατηγική και αυτό δεν είναι... Προ... προέρχεται από την κυρία Μογκερίνη την ίδια. Η κατάσταση δεν είναι business as usual, δεν είναι το σύνθε σενάριο. Βασιζόμαστε στην αναπτυξιακή πολιτική. Η, η κοινή γνώμη ε, τι, βλέπει τους ε, ανθρώπους ε, φεύγουν από την Ερυθρία γιατί έχει δικτατορία. Στο Μάλι ε, ε φεύγουν γιατί είναι φτωχοί. Αναποδογυρίζουν τα σκάφη στην Λαμπεντούζα, στη Μεσόγειο και ξαφνικά τότε Βλέπουν οι άνθρωποι αυτή την κατάσταση και κάποιοι ασχολούνται με αυτό το δράμα, άλλοι ασχολούνται με τη διαρθρωτική φτώχεια ή τη φτωχή διακυβέρνηση, την κακή διακυβέρνηση σε αυτά τα κρατημέλη ή ξέρω εγώ πλήττονται από το Ελληνίνιο ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε και είναι το πρόβλημα. Και ανακαλύπτουν ξαφνικά τον κόσμο, τι συμβαίνει. εντάξει υπάρχει η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινή γνώμη, αλλά από πλευρά πολιτικής πρέπει να υπάρχει μία διάρθρωση. Δεν δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα σε αυτή την τόσο μεγάλη κλίμακα με τις απώλειες ζώων και να πούμε ναι, αλλά αυτό ε, ταιριάζει με την επίσημη αναπτυξιακή μας βοήθεια, ODA. Τι σημαίνει αυτό πρέπει φυσικά να υπάρχει συμβατότητα, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ε, αυτά τα σχεδόν 2% να τα χάσουμε. Ε, και βάσει των εκθέσεων ε, και του το κανονισμού θα δράσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποκλίνουμε. Φυσικά όμως υπάρχουν ναι, και μονομένες δράσεις. Να το συζητήσουμε αυτό, αλλά το μόνο που κάνουμε είναι να είμαστε duckable, να συμφωνούμε με αυτή την πολιτική που έχουμε ε, αποφασίσει, ε, ε, δεν εκτρέπουμε τα, τα χρήματα. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι φέρουμε και μία ευθύνη ε, πρωτοβουλίες να καταθέσουμε προτάσεις και γι' αυτό προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτή την πρόκληση. Δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε να μοιράζουμε χρήματα με αυτόν τον ε, κατακαιρματισμένο τρόπο, διότι δεν είναι δίκαιο. Δεν ισχύει ότι ε, απέτυχε παταγωδός η αναπτυξιακή πολιτική και τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιοι ε, που βρίσκονται σε καλύτερη θέση και συνέβαλε σε αυτό η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτίμηση που έγινε για τους στόχους χιλιετίας ε, ήταν εν μέρη θετική. Δηλαδή όλοι συμβάλαμε και εν μέρη επιτύχαμε αυτούς τους αναπτυξιακούς στόχους. Είναι εν ο κόσμος και φυσικά μιλήσει Γι' αυτό σας έλεγα για την κινητικότητα, αλλά δεν μετακινούνται μόνο οι άνθρωποι, αλλά και στο εσωτερικό των φτωχών από στατιστικής ε, ε, κρατών υπάρχει μετακίνηση. Δηλαδή, ή μπορεί να είναι στατιστικός πόσο πλούσιες, αλλά να έχουν φτωχότερες περιοχές και μετακινούνται οι άνθρωποι στο εσωτερικό των χωρών. Θα πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτά τα φαινόμενα, δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή την, ε, αυτό το φαινόμενο της φτώχεια, με την κινητικότητα. Υπάρχει, ναι, και γι' αυτό είμαστε σε ένα σταυροδρόμιο, είναι σε καμπή η αναπτυξιακή μας πολιτική και Πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν, το θέμα δεν είναι να ε, μαλλιοτραβιόμαστε ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ναι, και είναι λίγο κατακαιρματισμένο, αλλά είναι να μπει στο επίκεντρο η μετανάστευση. Ταυτόχρονα όμως ε, να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες ε, που δικαίως ή αδίκως, αδίκως πιστεύω εγώ, ότι αυτό αυτή η απειλή αυτη η απειλη ειναι στο κέντρο των εξελίξεων. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση, όμως ξέρετε, αυτό το φαινόμενο ασκεί πολύ μεγάλη πίεση ε, στα θεσμικά όργανα για να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και κάποιοι πολλούν ακριβώς αυτή την ερμηνεία ότι είναι ανεξέλιγκτη η κατάσταση. Φυσικά υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν επιδοκιμάζω, αλλά ξαναλέω από πλευρά των εταίρων μα, αλλά ξαναλέω θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί μου. Δεν είναι δικό μα το πρόβλημα, είναι ε, πρόβλημα ολονών. Θα είμαι πιο συγκεκριμένο τώρα. Όταν προσδιορίζετε την αιρεσιμότητα, τι σημαίνει στην ουσία μέσα σε ένα διαστρωμένο διάλογο να δούμε πώ μπορούμε να συμφωνήσουμε σε επί πιθανών λύσεων. Αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, τι θα κάνουμε για να δούμε. Μέσα στο έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί Βλέπετε την πρόταση. Δεν υπάρχει στόχος να... Κανένα στόχο να τιμωρήσουμε κάποιον. Ακόμη και για κράτη που μπορεί να ισχυριστεί κάποιο ότι δεν τηρούνται τα πρότυπα τη ε, διακυβέρνηση. Ε, κάνουμε τη διάκριση και στην Ερυθρέα. Ξέρετε, έχει συζητηθεί επί πολλή και πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στου πολίτε ερυθρέα και την κυβέρνηση τη Ερυθρέα. Γιατί στοχεύουμε του ανθρώπου αυτέ τι συμφωνίε, ε, Γιατί θέλουμε στην ρίζα τη να τη χτυπήσουμε τη φτώχεια ναι, ε, πιεζόμαστε για την αναδεξιακή πολιτική, ναι είναι σε καμπή, γιατί καθημερινά οι πολιτέ αυτό μας ρωτάνε. Τι τα κάνετε τα 50 δις ε, για την αναδεξιακή πολιτική για τα 5 χρόνια του ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαίσιου. Δεν τα διαχειρίζομαι εγώ, εγώ είμαι ένας ταπεινός υπάλληλο, αλλά μας ρωτάνε τι τα κάνετε. Πρέπει να τους δώσουμε μια απάντηση. Για τη μετανάστευση να σου πούμε, Φερρυπίν, συγκεκριμένα αποφασίσαμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουμε τη μετανάστευση ως βασικό άξονα ε, της αναπτυξιακής πολιτικής. Μπορεί εσείς να το διαφωνήσετε, αλλά αυτή είναι η απάντηση που δώσαμε. Δεύτερον, είναι κάθετη η επιχείρηση και ας δεν ασχολούμαστε με τις βαθύτερες, ρίζες, τη φτώχεια κτλ. Όχι, σε καμία περίπτωση όμως πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνουν αυτές οι αιτίες. Κλιματικές αλλαγές, ε, φτώχεια, διαρθωτική φτώχεια, αστάθεια, ε, κακή διακυβέρνηση, πόλεμος ε, και ούτω καθεξής. Φυσικά με διαφορετικά μέσα θα τα αντιμετωπίσουμε αυτό, όχι μόνο με αυτά που σας προτείνουμε τώρα. Έχουμε μία πληθώρα μέσων, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας πρώτα πρώτα ότι η μετανάστευση και κινητικότητα που δημιουργεί και ευκαιρίε αλλά ταυτόχρονα και ε, πολλά βάσανα για πάρα πολλού ε, είναι πλέον στο πυρήνα τη αναπτυξιακή πολιτική. Τέταρτο. τι θα κάνουμε με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. 500 εκατομμύρια επιπρόσθετα κινητοποιούμε, να τα βάλουμε στο Trust Fund για να έχουμε τώρα ρευστό να κινηθούμε ξέρω, είπατε για τον έλεγχο, το δημοκρατικό έλεγχο. Ξέρετε τι απαντούμε συνήθως. Δημοσιεύουμε τις εκθέσεις, διαρκώς τα συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπουν κάπου αυτά τα κονδυλία για να διοχετευθούν άμεσα μετά από τη συζήτηση με του εταίρους μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να λάβουμε μέτρα. Σε καμία περίπτωση δεν χρηματοδοτούμε εμείς τις επιστροφές. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο. Δεν πληρώνουμε από κονδύλια ODA επίσημες αναπτυξιακή βοήθεια για να επιστρέφουν οι άνθρωποι. Και επίσης για το ρυθμό των επιστροφών, για το σχολιάσατε και αυτό, δεν είναι τόσο υψηλό. θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε αν ήταν διαφορετικός ο ρυθμός. Ούτε σεντ, ούτε τίποτα, ούτε δεκάρα τσακιστή δεν θα δώσουμε για τις επιστροφές. Και δεν Μπορώ εγώ να αποποιηθώ την ευθύνη για να σου πω ότι δεν είναι δική μου δουλειά. Μα θα, δεν, μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να τους βοηθήσουν, να καταλάβουν πρώτα απ' όλα. Ε, να, να, να καταλάβουμε κι εμείς από πού φεύγουν, πού πάνε. Γιατί ε, τα, τα λεφτά τελικά ε, έρχονται από την δεξιακή πολιτική. Πρέπει να ξέρετε, ε, και να ξέρουν ότι αυτό θα κάνουμε. δεν πληρώνουμε. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για τι επιστροφέ. Αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε. Συμφωνία επανεισδοχή. Έχουμε αυτό το άρθρο 13 τη Κοτονού. Δεν επιτρέπει τέτοιε συμφωνίε επανεισδοχή. Πολύ καλύτερα συμβαίνουν αυτά στα πλαίσια ενός διαλόγου παρά να αρχίσουμε με ατέρμονε ανεπίσημες διαπραγματεύσει. Επόμενο σημείο όσον αφορά τα κονδύλια. Μα τα περισσότερα, μεγαλύτερα, σημαντικότερα ποσά ήδη υπάρχουν. Χρησιμοποιούμε απλώς κάποια νέα χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις. Θα μπορούσα να σας απαριθμίσω πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε όσον αφορά τις νεώσιμες πηγές ενέργειας. Επενδύσεις για να δημιουργηθούν οικονομικές δραστηριότητες, θέσεις απασχόλησης. Εγώ αναφέρομαι στις κλασικές υποδομές και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα. Να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και αυτό το αναφέρουμε στην ανακοίνωση. Ήδη βλέπουμε ότι αυτή η δυνατότητα ανάμιξης πολλών διαφορετικών μέσων, blending, αποδίδει κάποια αποτελέσματα. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή επενδύσεις πολύ μεγάλης κλίμακας, αλλά έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε δημόσιους και ιδιωτικού πόρους. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό κατακαιρματισμένα αυτή τη στιγμή, πάντως το φθινόπωρο θα έχουμε μια νέα νομοθετική πρόταση, η οποία θα εγκριθεί μέσω της διαδικασία της συναπόφασης και η οποία θα αντιστοιχεί στο σχέδιο Juncker. Όπως είχαμε κάνει και με το επιδετικό σχέδιο Juncker, έτσι θα πρέπει να κάνουμε και μία συζήτηση για τα επιδετικά σχέδια της εξωτερικής μας ανεπτυξιακής πολιτικής. Θα μας δοθεί λοιπόν η δυνατότητα να κάνουμε μια ενδελεχή συζήτηση και για το ζήτημα αυτό, ένα εξωτερικό δηλαδή επενδυτικό σχέδιο. Τώρα, το ότι δίνουμε χρήματα και δεν έχουμε απτά αποτελέσματα. Μα δείτε για παράδειγμα τα αριθμητικά δεδομένα για την Τουρκία, την Ανατολική Οδό, τα Βαλκάνια. Έχοντας επενδύσει τώρα στην Τουρκία και το είχαμε κάνει και περισσότερο στο παρελθόν, οι επενδύσεις αυτές πάντως η χρηματοδότηση βοήθησαν στην αχέτηση των παράτυπων μορφών μετανάστευσης και βοήθησαν στη πάρα, διάσωση πάρα πολλών ζώων και καταφέραμε κατά αυτόν τον τρόπο να υποστηρίξουμε και την επανένταξη των ανθρώπων αυτών που επιστρέφουν στην Τουρκία. Επανένταξη στην αγορά εργασίας, επανένταξη στις κοινωνίες, Είδατε και τη δήλωση του Ερτογάν όσον αφορά το ζήτημα της υπηκότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει σαφής βελτίωση. Τώρα, όσον αφορά την κεντρική Μεσόγειο, αντιμετωπίζουμε τώρα μια κατάσταση και καταβάλουμε προσπάθειες για να σταθεροποιήσουμε τη Λιβύη. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επί του παρόντος όμω, προσπαθούμε να δούμε στη θάλασσα τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολλέ και στρατιωτικές αποστολές όπου σώσουμε περισσότερες ζωές, σαφώς περισσότερες από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές έχουμε καταφέρει να διασώσουμε. Πρέπει όμως να φτάσουμε μέχρι το Σαχέλ για να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μετανάστευσης. Γιατί σαφώς θα πρέπει όχι μόνο να σταματήσουμε τα δίκτυα παράνομης διακίνησης, αλλά να συνεργαστούμε με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, προκειμένου να καταφέρουμε να σταματήσουμε τις δράσεις αυτές. Και με, το, με την κυρία Βασιλιάδου μιλούσα πριν από πριν από μερικέ ε, μέρε, που είναι υπεύθυνοι για το ζήτημα αυτό, και είπε ότι ακριβώ με τι χώρε αυτέ τη Αφρική θα πρέπει να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουμε εκεί τι απαραίτητε ικανότητε, προκειμένου να μπορούν και αυτέ να μα βοηθήσουν στην αναχέτηση των μεταναστευτικών ροών και στην εξάρθρωση των δικτύων παράνομη διακίνηση. Διαφορετικά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και οι χώρε αυτέ, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι ελοχεύουν από την μη σωστή διαχείριση των συνόρων τους. Έχουμε τους 80.000 αυτούς πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται στην Αιθιοπία, από τη Σομαλία, την Ερυθρέα και από άλλες περιοχές. Αυτή τη στιγμή κινητοποιούμε πόρους προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε περισσότερο εκεί την κατάσταση, να καταφέρουμε να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς μια καλύτερη πρόσβαση στην κοινωνία, μια καλύτερη καλύτερε και πιο αξιοπρεπέ συνθήκε διαβίωση. Αυτό ήδη το κάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι λοιπόν να γίνεται αυτό όχι με τρόπο κατακαιρματισμένο, αλλά με τρόπο συντονισμένο και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Στόχος μας δεν είναι αυτή τη στιγμή να έχουμε μία, ένα κατακαιρματισμό των χρηματοδοτήσεων που θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε πολλά παράλληλα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να προσανατολίσουμε τρόπο συντονισμένο τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να λέμε ότι, κοιτάξτε, αυτή είναι η βασική μας κοινή στάση, αυτή είναι η κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε και μέσω των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά που είπατε για την κυριότητα, τον εστερνισμό. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να ταποκριθούμε και στο ζήτημα αυτό σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ενδεχομένω να μην τα καταφέρουμε, θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα πάρα πολλέ δυσκολίε. Ο πειρασμό από την πλευρά των εταίρων μα είναι να πούνε ότι ναι, πολύ ωραία, μπορούμε να αποφεληθούμε από τα σύμφωνα αυτά προκειμένου να λάβουμε περαιτέρω χρηματοδότηση. Ελοχεύει όντω ο κίνδυνο αυτό, μα για να τον αντιμετωπίσουμε χρειαζόμαστε μια συντονισμένη, ολοκληρωμένη στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά σα είπα μέσα σε άκρε απαντώντα στις ερωτήσει σα και στις παρατηρήσει σα, όταν θα, μάλλον πότε θα αρχίσουν να λειτουργούν τα σύμφωνα αυτά. Μας είχε απασχολήσει και αυτό. Θεωρώ ότι μετά το καλοκαίρι θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη ιδέα για τα σύμφωνα αυτά. Θα δούμε τι μορφή θα πάρουν. Εμείς δεν τα προσεγγίζουμε ως νομικά δεσμευτικές συμφωνίες, αλλά περισσότερο ως πλατφόρμες, προκειμένου να καταφέρουμε να συντονίσουμε τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διάλογο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει με τις χώρες εταίρους. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβαστούμε τις διαδικασίες που έχουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. και ο κύριος Μίπιτσα και η κυρία Μογκερίνη είναι σε θέση να έρθουν εδώ πέρα για να συζητήσουν περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό και παντώ κατά αυτόν τον τρόπο και στην ερώτηση την οποία θέσετε σε σχέση με τον έλεγχο που θα πρέπει να ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε εταίροι για να αλλάξουμε τα πράγματα, θα πρέπει πραγματικά να καταφέρουμε να συντονίσουμε καλύτερα και τη διοργανική μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Υποθέτω ότι η ιδέα υπάρχει, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά για να πάρει σάρκα και ωστά η πολιτική αυτή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς πρόγραμμα, πώς να το πω, είναι μια άμορφη μάζα. Καλά, θα δούμε το Σεπτέμβριο. Ε, όταν γυρίσουμε τι διακοπέ, θα μα πείτε. Όταν, όταν δούμε μια τέτοια συμφωνία τότε θα καταλάβουμε περί τίνο πρόκειται ακριβώ. ωραία. Κύριε Γενική Διευθυντά, πολλέ ερωτήσει σα κάναμε. Τώρα πάμε θερινέ διακοπέ, αλλά εσεί θα έχετε πολλή δουλειά μπροστά σα. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μα. Να τον ευχαριστήσουμε που μα ήρθε. Λοιπόν, γρήγορα πάμε στο σημείο 7. Το συγγνώμη από τον Brian Hayes, διότι πρόκειται για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καπολέμηση εμπορίας αγρίων ειδών πανίδας. Ήταν μεγάλο το θέμα το προηγούμενο, μας έφαγε περισσότερο χρόνο, λυπάμαι πολύ. Συνάδελφοι, αν φεύγετε, παρακαλώ, χωρίς πηγαδάκια και συζητήσεις, εκτός εθούσης αυτά. Μ' ακούτε, όσοι φεύγετε, παρακαλώ αποχωρείτε ησύχως. Ε, δεν θέλω να έχουμε υποσυνεδριάσεις εδώ. Εδώ μιλώ για όλους, και τους συντονιστές και λοιπούς. Θέλω να πάω στο σημείο 7. Είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, για το σχέδιο δράσης για ε, την καταπολέμηση των ειδών των αγριών αυτών. Συνδέεται με την ε, φτώχεια, με την αναπτυξιακή βοήθεια. Μπράιαν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω το λόγο. Όπως είπες, η έκθεση αυτή προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να φύγετε, φύγετε ησύχω. Θέλω να ακούσω τον εισηγητή. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έκθεση Επιτροπής, ε, έλεγα, περιβάλλοντος και εγώ γνωμοδοτώ. Το Φεβρουάριο Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έφερε την έκθεση αυτή και είναι καλή γιατί είναι τρεις διαφορετικοί τομείς που έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα ε, της εμπορίας των αγριών ειδών. Είναι τρεις πυλώνες που βασίζεται η έκθεση. Το πρώτο είναι η πρόληψη ολόκληρη, ένα ολόκληρο κεφάλαιο, με πολύ καλές ιδέες που έχουν να κάνουν με τη συνειδητοποίηση, με τους επιχειρηματίες, να μαθαίνουν ποια είναι ε, τα καθήκοντά τους και οι νομικές τους υποχρεώσεις και ιδιαίτερα για την διαφύλαξη της άγριας πανίδας. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την καλύτερη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και να ενημερώνεται ο κόσμο ότι έχει υποχρεώσεις όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνείς και όχι μόνο εμείς και τα κράτη-μέλη για να επιβάλλουν τον νόμο εκεί. Και το τρίτο, ο τρίτος έχει να κάνει με την ενίσχυση ε, και τη σύναψη παγκοσμίων συμμαχιών, δηλαδή με άλλες περιφέρειες του κόσμου να συνεργαζόμαστε, να καταδεικνύουμε το πρόβλημα και να κάνουμε κάτι για να το λύνουμε. Τώρα, κατά την άποψή μου, μπορούν να συνοψιστούν ως εξή ε, οι βελτιώσει στην έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η προστασία της άγριας πανίδας είναι πάρα πολύ σημαντική για τις κατατόπους ε, κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις περιφέρειες αυτές ε, και από πλευράς βιοπικιλότητας. Θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό σε όλες τις συστάσεις που κάνουμε ως Κοινοβούλιο. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η παράνομη δραστηριότητα ε, και όχι μόνο για τις ίδιες τις ε, κατατόπους κοινότητες με τη λαθροθυρία. Ε, ολόκληρα οικοσυστήματα απειλούνται, αλλά και η κοινωνία μας και θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Εδώ πρόκειται για εγκληματικά στοιχεία που είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένα, τα οποία έχουν και πολλά λεφτά γιατί είναι πολύ κερδοφόρα αυτή η μπίζνα, η παράνομη, έχει αναγνωριστεί περίπου ότι πρόκειται για 10 με 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίων ε, που αλλάζει χέρια κλιματιών. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη ε, ε, αυτή η δραστηριότητα, η παράνομη και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι οι οποίοι είναι και τελείως αδίστακτοι και θα χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο, θεμητό και αθέμητο. και ζητάμε από πολύ φτωχούς ανθρώπους να αντιταχθούν σε τέτοιους λαθροθύρες στην περιφέρειά τους χωρίς να τους δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζονται. Μα οι άλλοι είναι πανίσχυροι και αδίστακτοι και ε, οι φτωχοί άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι στην πρώτη γραμμή. Επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε πληροφορίες σε αυτό το τομέα και αν πραγματικά θέλουμε να εργαστούμε πολύ σκληρά για τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να οικοδομήσουμε στις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουμε και έχει να κάνει και με τη συλλογή προφοριών. Ε, το κάθε κράτος χωριστά μετά να τα μοιράζομαστε με τρόπο συντονισμένο. Και ε, επόμενη πρόταση που κάνω ε, στον Εθρεμπόριο Άγρια Πανίδα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται καλύτερα οι νόμοι. Τι να του κάνουμε του νόμου αν δεν εφαρμόζονται. Αν δεν βλέπει ο κόσμο ότι πίπτει και ράβδο. Θα συνεχίσουν το τροπάρι του. Υπάρχουν αρχέ επιβολή του νόμου στα κράτη-μέλη. Εκεί θα πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια, εκεί θα πρέπει να το καταλάβουν. Ότι ε, αστυνομικέ αρχέ, ε, υπηρεσίε πληροφοριών θα πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και με βάση το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό. Και είναι υποχρεωμένοι να τα παίρνουν σοβαρά υπόψη. Αυτά είναι τα πέντε σημεία λοιπόν ε, με τα οποία εμπλουτίζω πιστεύω την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Μέχρι την Τετάρτη μπορούν να καταθέσουν οι συνάδελφοι τροπολογίες και με χαρά να τις δω. Και την τελευταία μέρα του Αυγούστου, Λίντα, νομίζω ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ο Dear colleagues, Ευχαριστώ. Πρέπει να προστατεύσουμε την χλωρίδα και την ε, Πανίδα από το Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα από τη Λαθροθυρία. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να ηγηθούμε του αγώνα κατά της ε, λαθροθυρίας, ε, να λάβουμε ε, ισχυρότατη δράση για να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, για να συνεργαστούμε με τις τρίτες χώρες, για να ανατραπεί αυτή η αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Έχει σοβαρότητα επιπτώσει το φαινόμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για το ευζήν των χώριων κοινοτήτων που επηρεάζονται από την λαθροθυρία, από το παράνομο εμπόριο, ε, ε, ε, τίθεται κινδύνο τα οικοσυστήματα και ένοπλες ομάδες ε, που δρούν σε διεθνές επίπεδο ε, βλάπτουν έτσι ε, χώρες κοινότητες τον οικοτουρισμό και το καθεξής. Μεγενθείται το φαινόμενο της ελαθροθυρίας και ξεκάθαρα χρειαζόμαστε συντονισμένη τράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν την πανίδα τους, να, να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν ε, την ε, άγρια ζωή ε, και μην ξεχνάμε και τις αιτίε αυτού του φαινομένου. Ας, μην, ας προστατεύσουμε τη ζωή. Η άγρια ζωή είναι ζωή. Ας προστατεύσουμε τη ζωή και τα, ζώντα, τα όντα που έχουμε στη διάθεσή μας. Μαρία Ευχαριστώ πολύ. Τώρα λίγο εκπλήσωμαι εγώ <laughs> με τον τρόπο που μας παρουσιάζετε την έκθεση, λέει η κυρία Χόιμπουχ. Πολύ πιο αισιόδοξα και θετικά μας τα λέτε από ό,τι έχει γραφτεί. Για μένα η έκθεση είναι υπεραισιόδοξη γιατί το κυνήγι και ε, θα ήθελα και μια πρόταση για την καταπολέμηση της σύρας αγρίων ε, ειδών. Είπαμε θα πρέπει να προστατεύουμε τη χλωρίδα και την πανίδα αυτοί κυνηγάνε τα ζώα αυτά για να τα έχουν ως τρόπεα. Ε, ε πολλές φορές υπολογίζουμε ε, το κόστος και δεν σκεφτόμαστε ότι είναι απαραίτητο τμήμα της βιοπικιλότητας. Ε, ανήκουν στη χλωρίδα και την πανίδα. Δεν το λέει αυτό η έκθεση. Ε, γιατί οι βιότοποι αυτών των ζώων όλο και μειώνονται. Τα ίδια τα είδη αυτά εξαφανίζονται. Αλλά δεν τα κατονομάζουμε. Να πούμε ότι μιλάμε για το ορεινό καιρό, βρε παιδιά, για τον ελέφαντα. Γιατί δεν τα κατονομάζουμε αυτά τα είδη. Τι θα πει άγρια είδη. Γιατί τόσο γενικά και αόριστα. Και η γνωμοδότηση θα πρέπει να είναι πολύ πιο οξία στον τόνο της όταν πρόκειται για τη λαθροθυρία. Συγγνώμη. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη συνεργασία με τις κυβερνήσεις να πιέσουμε όπου οι κυβερνήσεις είναι ε, πολύ αδύναμες και διεφθαρμένες. Ακούσαμε ότι πρόκειται για λαθρεμπόριο με τέτοια είδη από άγρια ζώα και λαθρεμπόριο σημαίνει εγκληματικότητα, άρα και οργανωμένη. Mit Waffenhandel oder mit... Αυτό μπορεί κανείς να το συγκρίνει με λαθρεμπόριο όπλων ή ναρκωτικών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει πολύ πιο έντονη διεθνή συνεργασία εκατέρωθεν. Δηλαδή και από τις χώρες που αγοράζουν και από τις χώρες που πολλούν. Θα πρέπει ε, παντού να συνεργάζονται περισσότερο οι αστυνομικέ αρχές, τα δικαστήρια. Χρειαζόμαστε ανταλλαγή πληροφοριών για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ε, πραγματικά αποτελεσματικά. Και αυτά θα πρέπει να μπουν με πιο έντονο τρόπο στην γνωμοδότηση, έτσι και πιο όξη. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύντομα αν έχετε να πείτε τίποτα, κύριε Εμμανουέλ Μέρ. Σύντομα μόνο παρακαλώ. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, σας ευχαριστώ γιατί συμβάλλετε και εσείς στην όλη εργασία που γίνεται όσον αφορά το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών και επικεντρώνεστε στην ανθρώπινη διάσταση, σε αυτό το οποίο βιώνουν οι τοπικοί πληθυσμοί. Και ξέρετε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Be4 Life, ένα πρόγραμμα το οποίο ακριβώς με αυτή τη διάσταση ασχολείται επί τόπου και έχει ως στόχο να συμβάλλει στην συνύπαρξη τοπικών κοινοτήτων και άγριων απειλούμενων ειδών. Για μας ε, η αντιμετώπιση της ε, παράνομης εμπορίας άγρων ειδών, η καταπολέμησή της είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πρόβλημα είναι ότι ε, η παράνομη αυτή διακίνηση έχει πάρει παγκόσμια πλέον διάσταση, άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε και εμεί τα δίκτυα καταπολέμησης που έχουμε. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το ζήτημα της ζήτησης. Ζήτηση η οποία είναι πολύ υψηλή, ιδίω στην Ασία, και που τροφοδοτεί πάρα πολύ την παράνομη αυτή διακίνηση και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τη χρηστή διακυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κάνουμε όλη αυτή την εργασία στα πλαίσια του θεματολογίου 2030, στα πλαίσια των στόχων και συγκεκριμένα του στόχου 15-7, του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης που ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα της παράνομης εμπορίας ειδών λοιπόν μας απασχόλησε, το ζήτημα της λαθροφυρίας και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ζήτημα αυτό μας έχει απασχολήσει και στα πλαίσια της σύμβασης ΣΑΙΤΙΣ. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διεθνή αυτή σύμβαση όσον αφορά το εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη προτείνουν πλέον συγκεκριμένε κατευθυντήριε γραμμέ όσον αφορά το εμπόριο των τροπέων αυτών προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα όπου ακόμα και αυτού του είδους το κυνήγι για τα τρόπια θα διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες βιωσιμότητος ο εισηγητής παρακαλώ. Μα προσβλέπω αγαπητοί συνάδελφοι τις ε, τροπολογίες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Δύο σχόλια πρώτον. Υπόθηκε ήδη από ένα συνάδελφο ότι ε, είναι σημαντικό να δούμε ότι το ίδιο το κοινό έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες μας έχουν ζητήσει να πάρουμε περισσότερο στα σοβαρά το ζήτημα αυτό και να καταφέρουμε να αναλάβουμε δράσει σε διεθνέ επίπεδο για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε ενδιαφέρονται για το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει εμείς στην απάντηση που θα δώσουμε να λάβουμε υπόψη μας ακριβώς και τι ανησυχίε αυτές των Ευρωπαίων πολιτών. Δεύτερον, το ζήτημα των τρόπεων αναφέρθηκε σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαφώς θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, αν καταλήξουμε τελικά σε μια διεθνή συμφωνία η οποία θα μπορούσε να τροποποιηθεί προκειμένου να τονιστεί ότι όντως θα πρέπει να ληφθεί συγκεκριμένη δράση για το ζήτημα αυτό, τότε θα ήθελα όντως να το περιλάβω αυτό και στη δική μου την νομοδότηση. Και νομίζω ότι ε, δεν θα πρέπει να λέμε ότι δεν ασχολούμεθα με το ζήτημα της βιοπικιλότητος. Το αναφέρω και αυτό στην γνωμοδότηση, ότι όντω θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή, αλλά από την άλλη θα πρέπει και αυτές οι τοπικές κοινότητες να μπορούν να έχουν ένα βιώσιμο μέλλον, να μπορούν να είναι και στο μέλλον ευημερούσες κοινότητες. Προσβλέπω λοιπόν τις τροπολογίες που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι και όπως είπα και σε σένα Λίντα, Νομίζω ότι στις 31 Αυγούστου θα μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε τη γνωμοδότηση αυτή, έτσι δεν είναι. Ναι. Πέμπτη, 14 Ιουλίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και όντως θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Περάσουμε τώρα στο 8 της ημερήσιας διάταξης, γνωμοδότηση του κυρίου Ντέβα, ο οποίος είναι καθοδόν αυτή τη στιγμή Συζητάμε ουσιαστικά το προπολογισμό για το οικονομικό έτος 2017. Κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην προηγούμενη συνεδρίασή μας, όπου είχαμε τότε και τον εισηγητή από την Επιτροπή Προπολογισμών. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο προπολογισμού του 2017, αλλά με μια κάποια καθυστέρηση και αυτή τη στιγμή πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος για να καταφέρουμε να εγκρίνουμε αυτό το προπολογισμό. Ο δικός μας στόχος να καταφέρουμε να δούμε περισσότερο προσεκτικά τι γραμμέ του προπολογισμού που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πιέζουν πάρα πολύ, όπω για παράδειγμα πώ θα συμβάλλουμε στο νέο ταμείο για την Τουρκία, Turkey Facility, να δούμε επίση τι θα γίνει με το μηχανισμό αναπτυξιακή συνεργασία. Αν δούμε λίγο τα αριθμητικά δεδομένα, και ελπίζω ότι είναι καθοδόν ο κύριο Ντέβα, φαίνεται ότι το απόθεμα του μηχανισμού αναπτυξιακή συνεργασία έχει μειωθεί τελικά προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματο. Ελπίζω ότι θα καταφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει περισσότερε πληροφορίε προ αυτό. Αγαπητέ συνάδελφοι, έλεγα απλώ ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έλεγα ότι ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταφέρει να μα δώσει περισσότερε πληροφορίε για το πώ θα επηρεαστεί ο μηχανισμό αναπτυξιακή συνεργασία από τη συμφωνία που έχουμε συνάψει με την Τουρκία. Επίση, θα θέλαμε να γνωρίσουμε για ποιο λόγο ο προπολογισμό για ανθρωπιστική βοήθεια είναι χαμηλότερο από πέρυσι. Κάθε φορά που συναντιόμαστε με προσώπους από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, τους λέμε κάθε φορά και συμφωνούν και αυτοί ότι οι ανάγκες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Πάντως δίνω το λόγο στον κύριο Ντέβα. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου. Uh, Ξέρετε ήδη ότι είναι υποπίεση ο... όλοι, ο προπολογισμό και όλοι που προσπαθούν να κάνουν τόσα πολλά με τόσα ε, λίγα λεφτά. και νομίζω ότι είμαστε σε μία κατάσταση όπου ο Επίτροπος πρέπει να βρει από κάπου λεφτά που δεν έχει όμως. Ε, είναι, λειτουργεί υπό μεγάλη πίεση ε, και πραγματικά σας συμπονώ. Έχω καταθέσει τη γνωμοδότηση και υπάρχουν και τροπολογίες ε, όπως ξέρετε. Θέλω όμως να κάνω πιο γενικόλογα σχόλια. Ε, για χούς μόχλευσης ε, καταφέραμε να βρούμε κονδύλια. Τι θα γίνει, τι απαιτείται. Ε, χρειάζομαστε συνεργασία με την αγορά για διάφορους σκοπούς. Εγώ έχω βρει χρήματα ε, στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και τι χρειάζεται, δέουσα επιμελητία, έλεγχος, ένα business plan, επιχειρηματικό σχέδιο, έλεγχος αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου. Και όλα αυτά απαιτούν παρακολούθηση και έχω την εντύπωση ότι στην Επιτροπή ιδέα δεν έχουν από αυτά. Το θέμα λοιπόν είναι για το EDF και για το DCI πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις στάνταρ διαδικασίες που ε, ακολουθούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτήν τη χρηματοδότηση με μόχλευση. Θέλω η Επιτροπή να μας πει τι θα γίνει στη ΣΥΤΙ όπου θέλετε να αποταθείτε, πώς θα γίνει να συνεργαστούμε με αυτά τα χρυσά παιδιά για να έχουμε ε, τα χρήματα που χρειαζόμαστε για τη Δυτική Αφρική, για ε, μέρη του ε, εργαλείου για την ανάπτυξη, το DCI, όλα, δηλαδή όλα αυτή τη χρηματοδότηση μόχλευσης για να βρείτε αυτά τα 200-300 δίσε που θέλετε, πώς θα το κάνετε. Υπάρχει ένα το ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ξέρουν από αυτά εκείνοι. Αλλά περίεργος πώς δεν συζητούμε μαζί τους για αυτά τα ζητήματα. Το βρίσκω περίεργο αυτό. Θέλω να καταλάβω, να μου εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιο λόγο η ΕΤΕ δεν, δεν συνεργάζεται μαζί μας, αφού όμως έχει την τεχνογνωσία, έχει τις εμπειρίες. Ο Επίτροπος με παίρνει. Η Επίτροπος με παίρνει. Η Κρυσταλίνα. Κρυσταλίνα να σε πάρω σε δύο λεπτά. Γεια σου. Τώρα μιλάω στο κοινοβούλιο. Πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, καταφέρατε να σα πάρει η Κρυσταλίνα εκείνη ακριβώ τη στιγμή που μιλάτε στην Επιτροπή μας. Μας εντυπωσιάσατε. Λοιπόν, ε, από πλευράς λοιπόν χρηματοδότηση αυτά τα δύο θέλω να καταλάβω. Επίσης, θέλω η Επιτροπή να μας εξηγήσει ποια τμήματα της DCI που ελέγχει και το Κοινοβούλιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μόχλευση. για να μην δεν εξαρτώμαστε από τις χρηματοπιστωτικές αγορές μόνο, για να χρησιμοποιήσουμε στο DCI κάποιες γραμμές του προϋπολογισμού ως βασικό κεφάλαιο, το οποίο θα μοχλεύσουμε για να έχουμε πολλαπλασιασμό των κονδυλίων ε, που θα προέρχονται από τις επενδύσεις που θα κάνουμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τρίτον, έλεγχος. οικονομικός έλεγχος της ε, διαχείρισης αυτών των κεφαλαίων. Είναι πολλά τα χρήματα και όχι μόνο των φορολογουμένων αλλά και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Για το DCI χρειάζεται οικονομικός έλεγχος, τον έχουμε εν μέρη, αλλά για το EDF, για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, πλάκα μας κάνετε. Γιατί ε, υποτίθεται ότι έχουμε έλεγχο ε, μπορώ να σας πω και βάζω το, το, το, το, το ορκίζομαι επειδή ήμουν και στο Αγγλικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδέα δεν έχουν ναι, για πράγμα μιλάω από τη δική σας την εμπειρία Πόσα εθνικά κοινοβούλια ξέρουν τι τρέχει με το ε, Ταμείο ε, με το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και όταν μιλάμε για διαχείριση δισεκατομμυρίων, ποιο θα τα ελέγχει αυτά, ποιο θα, ε, θα είναι υπόλογο, ποιο θα, ποιος θα φέρει την ευθύνη. Κυρίε και κύριοι, μπορώ να σα πω, αν δεν έχουμε έλεγχο και απευθυνθούμε στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, δεν έχουμε σε επιμελητία και πάμε στη ΣΥΤΗ ή στη Φραγκφούρτη όπου θέλουμε να πάμε να βρούμε λεφτά, ξεχάστε το, αποκλείεται. Αν δεν θα μας δώσουν λεφτά, αν δεν έχουμε τις υποδομές απαιτούμενες για να κατοχυρωθεί ο έλεγχος, αν δεν χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες στάνταρ διαδικασίες των χρηματοπιστωτικών αγορών ε, που ακολουθεί οποιοδήποτε πάει να πάρει λεφτά από αυτές τις αγορές, δεν πρέπει να μας τα δώσουν. Και ε, θα πληγεί η αξιοπιστία της Ένωσης του και Ολονών, αν δεν κάνουμε τα μαθήματά μας πριν πάμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θα, πολύ θα ήθελα να μου απαντήσετε. Αν δεν ξέρετε, πείτε το. Ε, πείτε το. Ούτως ώστε να, βρούμε, ε, να βάλουμε μια τάξη ε, τους επόμενους μήνες. Για να πάω στα ειδικότερα σχόλια τώρα. Ζητάει η Επιτροπή μας από την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, σε αρμόδια Επιτροπή να σωματώσει ακούλουδε παρατηρήσεις στην πρώτη ψηφίσματος. Πρώτον, τονίζει ότι το φιλόδοξο θεματολόγιο 2030 ε, και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που συμφώνησαν το Σεπτέμβριο του 2015 τα κράτη-μέλη με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από απαιτούν ότι θα τηρηθούν τα επίπεδα του πολιετού σε δημοσιονομικού πλαισίου ενώ ε, διατηρούνται και οι μακροπρόθεσμες στόχοι του άρθρου 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την εγκλήρωση της στόχης. Δύο. Καλή από την Ευρωπαϊκή... Το έχουμε, το έχουμε το κείμενο. Το έχετε το κείμενο. Δεν χρειάζεται να μας το διαβάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, κυρία Εύες. Αυτά, αυτά, αυτές είναι οι προτάσεις που κάνουμε. είναι οι τροπολογίε που θέλουμε να υποβάλουμε να συμπεριληφθούν από την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα που πρέπει να θέσουμε. Τι κάνουμε με το Αφγανιστάν. για τις ε, ανάληψη που χρεώσουν για το Αφγανιστάν, αφού υποτίθεται ότι έχουμε κάνει και προγραμματισμό. Λέμε λοιπόν στην ε, γραμμή του προϋπολογισμού για την ανάπτυξη, έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια και εξαφανίστηκαν κάπου σε μια τρύπα 18 εκατομμύρια. Όμω κάνω λάθος, διορθώστε με. Η γραμμή για την ανθρωπιστική τώρα βοήθεια. 66,9 εκατομμύρια. Και 339 αντίστοιχα για το μέλλον. Χάθηκαν και αυτά. Πού πήγαν. Γιατί. Έχω γράψει και άλλα νούμερα, θα σας τα πω. Συνεργασία με την Ασία. Τι εννοούμε να το ξεχνάμε, θα είναι βασικός μας οικονομικός εταίρος. Και κάποιες χώρες ασιατικές θα χρειαστούν υποστήριξη. Μπαγκλαντές. και θα γίνουν πιο σημαντικές από άλλες ε, μουσουλμανικές χώρες. Άμα δεν παρακολουθείτε τις εξελίξεις ε, θα, θα, θα χάσουμε το τρένο. Γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Έχω και άλλες παρατηρήσεις. Θα σας τη στείλω γραπτός. Ναι. Και στην Επιτροπή και στην άλλη Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή. Θα σταματήσω. Θα σταματήσω γιατί αλλιώς δεν με σταματάει τίποτα. Ναι, έχουμε όλοι τα επτά σημεία, το σχέδιο νομοδότηση, το έγγραφο, όλα κομπλέ. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που λέτε και πολύ καλά σας κατανοούμε. Ο κύριο Λίτς έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ναι, θα έχει κάνει τροπολογίες για τους πρόσφυγες και την εκπαίδευση των παιδιών του. Ο κύριος Λίτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, να τις τα πείτε στο τηλεφώνημα που θα ακολουθήσει αυτά που θα σας πω. Λοιπόν, γενικώ ε, καλωσορίζουμε την αύξηση της ανάληψης υποχρεώσεων στο DCI το 2017. Ε, θα ήθελα όμως να τονίσω τα εξή δύο που θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο. Μειώνονται οι πιστός πληρωμών στην κατηγορία 4 από τη μια κατανοώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα ε, του προπολογισμού 2016, όπου χρειάστηκε να πληρώσουμε πάρα πολλούς καθυστερημένους λογαριασμούς προηγουμένων ετών. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος τώρα να ξαναδούμε την κατάσταση του 2015. Μειώνοντας τις πιστώσεις πληρωμών δηλαδή, δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις αναλήψεις υποχρεώσεων μας. Άρα, θα πρέπει να επανέλθουν οι πληρωμές ε, στο επίπεδο της ανάληψη υποχρεώσεων. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεύτερον, ε, η μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας. Το είπατε και πριν, Λίντα. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτε έχουμε θέμα με αυτό, ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι πληρωμές περικόπτονται ριζικά. Κανονικά θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο. Ε, να έχουμε αναπτυξιακή, ε, ανθρωπιστική βοήθεια και επιστημιστική με βάση τις ανάγκες και την τρέχουσα κατάσταση. Δεν μπορούμε τώρα λοιπόν να μειώνουμε παντού όλα αυτά τα κονδύλια γιατί είναι οξία η κατάσταση και τα προβλήματα πολύ σοβαρά. Ιδιαίτερα πέρυσι ε, δεσμευθήκαμε να βάλουμε 26 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια στην εκπαίδευση στους καταβλισμούς των προσφύγων. Ε, Εντούκα λέγεται η πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και θα παραμείνει η προτεραιότητά μας και για το 2017 και θα πρέπει να το μελετήσουμε και τα επόμενα χρόνια να το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Η Μαρία Χόιμπουχ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Äh, ε, μαζικές ε, μεταφορές πιστώσεων σε σχέση με το 2015 και έχουν μειωθεί και, τα, και έχουν κοστεί οι περικοπές και τα προγράμματα ε, θα πρέπει οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν για να καταργηθούν αυτές οι περικοπές για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, ασκεί μαζικότατη κριτική ο κύριος Ντέβα ότι έχει περικοπεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει μα, ότι είμαστε σε ένα κανονικό επίπεδο πάλι. Παρ' όλα αυτά παραμένουν ζητήματα και ερωτηματικά και συμφωνούμε μαζί σας μέσα προς το εξή. Οι προτάσεις ε, ε, που γίνονται ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και τα χρήματα πηγαίνουν, απορροφώνται από πραγματικές ανάγκες. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ρωτήσει, να μας απαντήσει και να την πιέσουμε εμείς αυτό. Και ένα τελευταίο έχει να κάνει με τις μεταφορές πιστώσεων που έχουν να κάνουν με την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, εκεί παίρνουν λεφτά και τα χρησιμοποιούν για την Τουρκία, όπως και για το Αφγανιστάν. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί το κάνουμε αυτό. Παίρνουμε λεφτά από φτωχές ασιατικές χώρες που χρειάζονται πηγόντως την αναπτυξιακή βοήθεια και τη δική μας χρηματοδότηση για να τα δώσουμε στην Τουρκία και το Αφγανιστάν διότι αυτό είναι προς όφελος των ε, τελείως ιδίων μας συμφερόντων. Είναι ιδιοτελής αυτή η αναπτυξιακή πολιτική και μάλιστα από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάμε δηλαδή τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της καταπολέμησης στόχης και της συνεργασίας. Θα πρέπει να τα πούμε αυτά έτσι με πολύ επικριτικό μάτι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άικ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, δεν ξέρω αν θέλουν άλλοι συνάδελφοι. Παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να μιλήσω για τον προϋπολογισμό του 2017. Όπως γνωρίζετε είναι πάρα πολύ δύσκολος και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα διάφορα ερωτήματά σας. Πρώτον, πώς το DCI συνεισφέρει ε, στη διευκόλυνση για την Τουρκία. Ε, ναι, είναι γεγονός αυτό. 115 εκατομμύρια πήραμε από εκεί για να τα δώσουμε στη διευκόλυνση της Τουρκίας και τα χρήματα αυτά προέρχονται κυρίως από αποθεματικά ε, προγραμματισμένα γεωγραφικές πραγματικές περιοχές αυτές, κυρίως Λατινική Αμερική και Ασία, που καλύπτει το μέσον DCI. Δυστυχώ μόνο αυτά τα κονδύλια υπήρχαν για από εκεί μπορούσε κανεί να τα αντλήσει. Εξού και έγινε αυτό. Γι' αυτό και βλέπετε να υπάρχουν διάφορες μετακινήσεις από τις διάφορες γραμμές. Έχουμε και front loading και back loading, δηλαδή και μπροστοβαρείς ε, ε, χρηματοδοτήσεις, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να τηρήσουμε ε, τον προγραμματισμό του μέσω στον DCI, αλλά ανάλογα με την οριμότητα των έργων και τις επίγουσες καταστάσεις, προσπαθούμε και εμείς να κανονίσουμε την πορεία μας και να κατανέμουμε διαφορετικά τα κονδύλια από χρόνο σε χρόνο. Αυτό είναι κυρίως το ζήτημα. ανησυχείτε για την Ασία και το Αφγανιστάν κυρίως. Σήμερα το πρωί είδα την πρώτη πρόταση του Συμβουλίου και νομίζω ότι συνεδριάζουν αυτή τη στιγμή με τη Γενική Διεύθυνση ε, Προϋπολογισμού. Όντως το Συμβούλιο έχει αρχίσει να κάνει τις πρώτες περικοπές που είναι 60 εκατομμύρια για το κεφάλαιο 4 εκ των οποίων 50 για τα κονδύλια και τις γραμμές ε, από την ΤΕΦΚΟ. 9,4 εκατομμύρια, Αφγανιστάν 5 από την Ασία, 10 εκατομμύρια από το μέσο για την Αφρική, το Παναφρικανικό συγκεκριμένα. 10 εκατομμύρια επίσης για τη Λατινική Αμερική και κάποιες άλλες περικοπές ε, για το περιβάλλον και την επιστηστική ασφάλεια. Και όντως έχει σημασία. Και παρακαλώ την Επιτροπή σας, απευθύνω έκκληση, να μας βοηθήσετε να ε, μην περάσουν αυτές οι περικοπές, γιατί θα είναι δραματική η κατάσταση, αν γίνει κάτι τέτοιο. Για το Αφγανιστάν. Σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, τι διαφορά υπάρχει. Αυξήθηκε η διαθεσιμότητα και είχαμε ένα backloading για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Ε, το άλλο που αναφέρατε είναι ε, is και το blending, δηλαδή η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και συνένωση πόρων. Και στην Ασία και στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική ε, υπάρχουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί. Λειτουργούν καλά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν αποκλείεται καθόλου. Συμμετέχει, αλλά δεν είναι ο αποκλειστικό εταίρος. Υπάρχουν και άλλες αναπτυξιακές τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω ότι είναι κάτι που λειτουργεί πολύ καλά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια που είναι βασικός τομέας. Υπάρχει πρωτοβουλία Electrify για τον εξελικτρισμό. Είναι 20 τα έργα που έχουν επιλεγεί και αρχίζει η χρηματοδότησή τους και η λειτουργία τους. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, έχει στηθεί καλά. και συνεργαζόμαστε με αυτές τις τράπεζες έτσι ώστε να βρεθούν τα κονδύλια και να ε, χρηματοδοτηθούν τα έργα. Κύριε Ντέβα, όταν είπατε ότι η Βουλή Βρετανική δεν ασχολείται ε, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, εγώ κάθε φορά που πηγαίνω στο Συμβούλιο και υπάρχει σκρούτινη reserve των Βρετανών, γιατί θέλουν να το περάσουν από το κοινοβούλιο τους. Γιατί ε, ακριβώς περνάει από το κοινοβούλιο. Εδώ πρόκειται περί διάσταση απόψεων. Δεν ξέρω εσωτερικά πώς είναι οι διαδικασίες στη Βρετανική Βουλή, αλλά είναι οι μόνοι που πάντα προβάλλουν αυτή την επιφύλαξη μελέτης από πλευρά του Κοινοβουλίου τους όταν ζητούμε κονδύλια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη. Έρχομαι τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τις πιστώσεις πληρωμών Όντως φέτος είναι έτος ρεκόρ ως προς τις πιστώσεις πληρωμών για τον απλούστατο λόγο ότι βγαίνουμε από, έξι, ε, από τρία χρόνια συγγνώμη, ελλείμματος. <clears throat> Πρόπερση η ΔΕΦΚΟ έκλεισε με ένα έλλειμμα περίπου 700 εκατομμυρίων στο τέλος του έτους Δηλαδή αυτά ήταν ε, ανεξόφλητοι λογαριασμοί και τιμολόγια που έπρεπε να πληρωθούν από τον προπολογισμό του 2015. Το 2015 κλείσαμε με άλλο έλλειμμα και πάλι 500 εκατομμύρια περίπου. Οπότε καταλαβαίνετε και φέτος ε, και πάλι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση περίπου σταθερή και πληρώσαμε ήδη 1,5 δισεκατομμύριο. Δηλαδή περίπου είμαστε στο 50% των υποχρεώσεών μας ε, των καθιστουρμένων πληρωμών. Δυσκολίες δεν προβλέπονται φυσικά. Φέτος έχουμε αρκετά χρήματα, ούτε του χρόνου. Και επειδή δεν θα υπάρξει λοιπόν ε, τεράστιο αυτό ποσό μισό δισεκατομμύριο μεταφορά για να πληρώσουμε του χρόνου, με τις πιστώσεις που ζητάμε νομίζουμε ότι είμαστε ρεαλιστικοί στην προσέγγιση μας και δεν θα έχουμε την κατάσταση το 13 στο 15. Ελπίζω να απάντησα σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντέβα, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, μα μου κάνει εντύπωση, πραγματική εντύπωση, η τελευταία αυτή δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα αιματηρή θα έλεγα ότι ήταν έτσι πολύ κοινική όσον αφορά τα ταμεία αυτά στα οποία αναφέρθηκε, τα κονδύλια στα οποία αναφέρθηκε. Για ποιο λόγο πιστεύετε πραγματικά ότι θα έχουμε τα χρήματα αυτά και ότι θα γίνουν οι πληρωμές. Μας λένε ότι έχετε ακόμα πάρα πολλές υποχρεώσεις όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και ότι εκεί προβλέπονται πολύ σημαντικές περικοπές. Πιστεύετε, εσείς μας λέτε ότι δεν θα έχετε έλλειμμα. Δεν έχουμε όμως κανέναν από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ αυτή τη στιγμή για να μας μιλήσει για την ανθρωπιστική βοήθεια, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ που θα μπορούσε να μας διαφωτίσει όσον αφορά τα δημοσιονομικά ζητήματα. Πολύ ωραία. Τελευταίο ερώτημα και θα περάσουμε στην έκθεση του κύριου Νόιζερ. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα το οποίο απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θα πρέπει να ενημερώσουμε τον αρμόδιο επίτροπο. Για ποιο λόγο άλλωστε δεν είναι εδώ πέρα κάποιο εκπρόσωπο από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Το ζήτημα της χρηματοδότησης ανθρωπιστικής βοήθειας είναι κρισιμότατο ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αποκριθούμε στι υποχρεώσει μα και να έχουμε και τι απαραίτητε πιστώσει πληρωμών. Ε, ναι, ενδεχομένω θα μπορούσαμε να βάλουμε όλα αυτά τα χρήματα σε κάποιο απόθυμα, λέει ο κύριο Δέβε, και να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, η 9η Αυγούστου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στη συνέχεια στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 31 Αυγούστου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την καθυστερημένη έγκριση του σχεδίου προπολογισμού, καθώς επίσης και την τοποθέτηση του Συμβουλίου, η Γραμματεία μπορεί να αποδεχθεί και οριζόντιες τροπολογίες, αν επιθυμείτε να υποβάλλετε τροπολογίες πριν την τοποθέτηση του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη δράση όσον αφορά τις διάφορες γραμμές του προπολογισμού, περιμένοντας βέβαια να δούμε και ποιες θα είναι οι προτινόμενες περικοπές από το Συμβούλιο. Στις 20 Ιουλίου συγκεκριμένα το Συμβούλιο θα καταλήξει σε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2020. Τι θα γίνει δηλαδή μετά την Κοτονού. Ξέρω ότι έγινε και μια συζήτηση στην προηγούμενη συνεδρίασή μας για το ζήτημα αυτό, γιατί εκείνη τη μέρα βέβαια είχαμε το δημοψήφισμα, δεν μπόρεσα εγώ να έρθω στην συνεδρίασή μας. Ο Νόμπερτ Νόιζερ είναι ο εισηγητή μα. Είχαμε 214 τροπολογίε. Επεξεργάζεστε, Νόμπερτ, αν δεν κάνω λάθο, κάποιε συμβαστικέ προτάσει αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσατε να μα σκεγγραφήσετε λίγο την πρότασή σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ja vielen... Ευχαριστώ. Ah. Äh, ευχαριστώ πολύ, Λίνα. Η έκθεση αυτή πιστεύω για την ε, μελλοντική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλά αναπτυσσόμενα κράτη, ιδιαίτερα με τις 79 χώρες ΑΚΕ, έχει ιδιαίτερη σημασία. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, τι θα γίνει μετά το Κοτονού σε πιθανή νέα συνθήκη, αυτό παραμένει ανοιχτό. Αλλά εμείς ως Κοινοβούλιο κάνουμε τις προτάσεις μας, δίνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές, είμαστε οι πρώτοι που τοποθετούμεθα και πιστεύω έτσι ότι ακριβώς επειδή πολύ νωρίς ασχοληθήκαμε με το θέμα μπορούμε να ηγηθούμε και στην επόμενη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με θετικό τρόπο να τα επηρεάσουμε. Δεν περί αυτολογώ, ούτε προσπαθώ να αποκτήσω την εύνοια των συναδέλφων, αλλά πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τους Κιώδης, τον Μωρίς Πονγκά, τη Μαρία Χόιμπουχ και το Λουί Μισελ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ γόνιμη η συνεργασία μας και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω από την ομάδα μας το Γέσπερ και το Ρενό για την καταπληκτική συνεργασία μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τις πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που μας ε, βοήθησαν πάρα πολύ και βεβαίως την Ολλανδική Προεδρία ακόμα και αν σε πολλούς τομείς δεν είχαμε πάντα ταύτιση απόψεων. Για τη δική μας έκθεση όμως ήταν πραγματικά σημαντικό και γόνιμο. Για να παραμείνει η έκθεση σε ένα ευανάγνωστο πλαίσιο, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε επαναλήψεις και επικαλύψεις και αυτό και τα βγάλαμε από τις τροπολογίες και νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά στις συμβαστικές προτάσεις, να τα συνοψίσουμε. Παραμείναμε πιστοί στη γραμμή μας, επικεντρωθήκαμε στα σημαντικότερα. Στο κέντρο, στον πυρήνα της έκθεσης είναι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε το πλαίσιο της συνεργασίας τύπου ΟΚΕ ο μεγάλος αριθμός χωρών είναι αδιαφυσβήτητο πλεονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα ε, ε, προσφέρει ποικιλία και ε, διαφορετικότητα και στο παρελθόν αυτό βάρινε και επιβράδυνε πολύ τη συνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν να προτείνουμε μια αρχιτεκτονική δομή για το μέλλον που να ενισχύει τη συνοχή αλλά ταυτόχρονα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα για να καλύψουμε λοιπόν και τους δύο αυτούς στόχους, τι προτείνουμε από τη μια και νομίζω μας έχει ε, είχε ο συμβιβασμό αυτός να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο για την συμφωνία για το τι θα διαδειχθεί το κότονου ε, και να κυριαρχούν στόχοι όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου ε, και στα πλαίσια αυτού να έχουμε πυλώνες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων περιφερειών και κρατών. <clears throat> Και να καλύπτεται έτσι και το καθημερινό πλαίσιο. Η πολιτική εταιρική σχέση αλλά και η κοινοβουλευτική διάσταση έχει για μας σημασία. Και στο μέλλον θέλουμε μαζί με τις χώρες ΑΚΕ να ε, φτάσουμε σε κοινούς στόχους με διεθνή παρουσία στα Ηνωμένα Έθνη ε, και στις διάφορες ε, συσκέψεις ε, δωρητών. Οι σχέσεις μας δεν θα πρέπει να είναι σχέσεις δωρητών και δικαιούχων, αλλά είναι επίσης όρις και με εταιρικό πνεύμα με βάση τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θελήσαμε να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει περισσότερο, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και στις χώρες ΑΚΕ ιδιαίτερα να ακούγονται περισσότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι ανάγκες έχει ο κόσμος ε, και πώς θα αποκρινόμαστε σε αυτά. Επί της ουσίας βασιζόμαστε στους στόχους ε, βιωσιμότητας, τους ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Ένα σημείο κριτική στη σημερινή συμφωνία είναι ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε σε πολλές χώρες την κατάσταση αυτή να βελτιωθούν και προτείνουμε να γίνεται έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναδιετία για να παρακολουθούμε την κατάσταση και όταν υπάρχουν παραβιάσεις να προειδοποιούμε αλλά και ταυτόχρονα να επιβραπεύουμε θετικές εξελίξεις στα ε, ε, κράτη αυτά με τα οποία συνεργαζόμαστε. <clears throat> Καλές εμπορικές σχέσεις είναι πάντα η βάση για τη συνεργασία, για να υποστηρίζουμε τις χώρες εταίρους μας, για να γίνουν ε, οικονομικά ανεξάρτητα και να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης του κόσμου. Αυτό για να λειτουργήσει χρειάζεται το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό περιβάλλον πραγματικά και το κλίμα να είναι πρόσφορο. Θέλουμε ε, να υπάρχουν πρότυπα ε, δεσμευτικά σε μια νέα συμφωνία τύπου ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αντίστοιχε αναφορές. Για το θέμα της συμπερίληψης ασφάλειας και ανάπτυξη στο τέλος κάναμε κάποιες συζητήσεις. Χρειάζεται σαφής διάκριση ανάμεσα σε αυτό που νοείται αναπτυξιακή συνεργασία για την καταπολέμηση της φτώχειας και την ασφάλεια. Γι' αυτό επιλέξαμε τη διατύπωση που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, σαφήνεια και συνοχή. Νομίζω σε αυτό, με αυτό το συμβασμό μπορεί να συμφωνήσουν περισσότερες πολιτικές ομάδες. Πέρα από όλα αυτά και χρονικά μετά την έγκριση της έκθεσης στην Επιτροπή που θα πάει στην Ολομέλεια ε, θα έχουμε λάβει εμείς θέση, καλή πιστεύω και θα περιμένουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που νομίζω ότι θα είναι σχετικά κοντά στο δικό μας αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα εναπόκειται σε εμά το πώς μπορούμε να τα περάσουμε όλα αυτά στα κράτη-μέλη. Θα είναι σκληρή αντιπαράθεση. Γιατί τον τελικό λόγο τον έχουν εκείνοι και αυτοί θα καθορίσουν. Και πώς πήγε η συνεργασία μας με τα 78-79 κράτη και, και πώς θα συνεργαστούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν για την έκθεση και τους συμβιβασμού και περιμένω με χαρά την ψηφοφορία μετά τις θερινές διακοπές. Με το καλό. Σα um, Σας ευχαριστώ, κύριος Πόγκα. Ευχαριστώ. Ε, αυτά που είπε ο εισηγητής. Ε, ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας. Θα ήθελα να το συγχαρώ για τη δουλειά που έκανε. Είμαι πεπισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσει αυτή την προνομιακή σχέση με τι χώρε ΑΚΕ. Όμω πρέπει να καταστεί αποτελεσματικότερη η σχέση για να ανταπεξέλθουμε στι παγκόσμιε προκλήσει. Α, και κάτι άλλο που μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα υπερπόδια διαμερίσματα που ε, έχουν τα ίδια μέσα προς το παρόν με τις χώρες ΑΚΕ θα έχουν ξεχωριστό ε, χρηματοδοτικό μέσο. Είναι πολύ διαφορετικό το πλαίσιο σε σχέση με τις χώρες ΑΚΕ και θα πρέπει να ε, προωθήσουμε και να τονίσουμε τις ιδιαιτερότητες που ισχύουν για αυτές τις χώρες. Μαρία ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και σένα Νόρμπερτ. Πολύ καλή δουλειά πραγματικά και εκ των προτέρων ε, συνεργάστηκες με όλους τους σκιώδεις και με μεγάλη ευρία διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων. Πάρα πολύ μας βοήθησε αυτό και σε ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση ε, πραγματικά σε λεπτομέρειες αναφέρεται στη μορφή συνεργασίας που επιδιώκουμε να έχουμε με τις χώρες αυτές μετά από πέντε χρόνια αλλά κατά την άποψή μου και ο εισηγητής αλλά και η Επιτροπή μας δεσμεύονται πολύ νωρίς για συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ακόμα δεν έχουμε την αξιολόγηση της Συμφωνίας Κοτονού, ε, τον απολογισμό δηλαδή. Και υπάρχουν διάφορα σενάρια και μορφές συνεργασίας, τα οποία δεν τα έχουμε σκεφτεί ακόμα, ούτε τα συζητούμε ε, επί της ουσίας. Υπάρχουν κάποιες ιδέες, έτσι, κάποια περιγράμματα, αλλά δεν έχουμε μπει σε λεπτομέρειες και δεν μπορούμε πολύ γρήγορα να ε, δεσμευτούμε για κάτι. Ε, το συζητήσαμε λοιπόν με τους κοιόδης συγητές για να δούμε τι μορφή στο μέλλον μπορεί να λάβει η συνεργασία έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός ο τρόπος λειτουργίας και να πιάνει τόπο. Αυτή η φόρμουλα και δηλαδή Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός, συν ε, κάποια παρένθεση, αυτό να είναι μια συνολική μορφή, είναι το καλύτερο. Ακόμα δεν μπορούμε αυτά να τα αξιολογήσουμε, να τα εκτιμήσουμε. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα υπάρχουν επικαλύψεις και οι αδυναμίες της συμφωνίας του Κοτονού δεν ανταπο... αντιμετωπίζονται μάλλον αποτελεσματικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. ασφάλεια. Στην Αφρική αυτό είναι αρμοδιότητα της Αφρικανικής Ένωσης, αφέστατα. Και εάν ε, συνεχίσει να υπάρχει ΑΚΕ, δεν ξέρω αυτό τι νόημα θα έχει και ποια προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι αρμοδιότητα λοιπόν της Αφρικανικής Ένωσης και όχι ΑΚΕ. Ε, ξέρω εγώ, αυτό είναι σκόπιμο. Περιμένω να γίνει σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση της Συμφωνίας ε, Κοτονού ε, που θα έρθει να επιβεβαιώσει μάλλον αυτό που λένε οι σημερινές αναλύσεις, ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες, ε, πολιτική συνεργασία, ε, εμπόριο και η τρίτη είναι αναπτυξιακή συνεργασία και από τους τρεις πυλώνες ουσιαστικά μόνο ο τρίτος λειτουργεί. Η αναπτυξιακή, οι χώρες και συνδέονται τεχνητά. Δηλαδή, μάλλον η ιστορική σύνδεσή τους είναι τελείως διαφορετικές. Ούτε κοινά συμφέροντα έχουν, ούτε κοινά προβλήματα. Και στο διεθνέ στερέωμα δεν έχουν ε, αναπτύξει αρκετά ισχυρή κοινή παρουσία. Οι δε διαφορετικές ε, περιφέρειες αυτές δεν έχουν κοινή προσέγγιση στη ε, διάδρασή τους και στο εμπόριο με ε, τη συνεργασία τους. Παράδειγμα, ε, η μετανάστευση. Η Συμφωνία Κοτονού προβλέπει εδώ διάλογο, αλλά όποιος ήταν στη ποιος ήταν παρόν στη Βαλέτα ε, τον Νοέμβριο, Αφρικανική Ένωση και όχι χώρες ΑΚΕ. Και καλά ήταν και σκόπιμο, γιατί αυτό το πρόβλημα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση και όχι τις χώρες ΑΚΕ στο σύνολό τους. Έχω λοιπόν τροπολογίες που ανταποκρίνεται και λαμβάνουμε υπόψη στα συμπεράσματα των ερευνητικών Ινστιτούτων και ζητώ να μην δεσμευτούμε τόσο πολύ, τόσο νωρίς. Παίρνω απόσταση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Συζητούμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ, ενώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι η Μεγάλη Βρετανία. Το ανέφερε η Λίντα Προηγουμένως είπε ότι είναι μια ανίποτη ε, απόφαση, εν πάση και ε, καθώς μας ε, αφήνει χρόνους η Μεγάλη Βρετανία, εμείς συζητάμε αυτή την έκθεση τώρα για τις σχέσεις μας με τις χώρες και για την αναπτυξιακή συνεργασία και για την εμπορική πολιτική. Η Τανζανία αποφάσισε να μην υπογράψει τη σχέσεις εταιρικής και μάλλον οικονομικής τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Πολύ νωρίς είναι λοιπόν για να δεσμευθούμε. Περιμένετε να δούμε τι θα διαδεχθεί τη Συμφωνία Κοτονού. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, I think we need to... Ναι, Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και ποιο θα ο αντίκτυπο τη απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πολύ νωρί αυτή τη στιγμή ακόμα. Πολλέ πτυχέ πρέπει να εξετάσουμε και δεχομένω οι συντονιστέ να πρέπει να διεξάγουν μια συζήτηση το φθινόπωρο για τα διαφορετικά ζητήματα τα οποία θα θυγούν, όπω αυτέ οι εταιρικέ σχέσει στι οποίε αναφερθήκατε. Μέχρι την Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε νέα πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα Πρωθυπουργό, Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το όνομα αυτής Τερίζα Μέη. Εδεχομένω λοιπόν να αρχίσει να αποσαφηνίζεται η κατάσταση πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Λόλα Σάντζε. Ευχαριστώ Λίντα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νόησερ για τη δουλειά που έχει κάνει. Παρόλο που πιστεύουμε και εμεί ότι η Επιτροπή μα εδώ θα πρέπει να ποντάρει ε, σε ένα μέλλον σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης που να βασίζεται σε μια εταιρική σχέση μεταξύ ίσων. Θα πρέπει να τερματιστούν οι απικιακές λογικές που σήμερα έχουν γίνει ασήμαντρες οικονομικές σχέσεις με ένα νέο είδος απικιοκρατίας οικονομικής. Θα πρέπει να έχουμε αμοιβαίο σεβασμό, αλληλεγγύη των λαών και συνεργασία. Με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κέντρο με τρόπο αποτελεσματικό, που πάει να πει δεσμευτικό, αλλιώς τι να τα κάνουμε. Πού είναι η αξιοπρέπεια του κόσμου. Θα πρέπει να κυριαρχεί στην εταιρική σχέση πάνω από εμπορικά συμφέροντα ολίγων. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς. Οι στόχοι των τριών διαφορετικών ε, πυλώνων θα πρέπει να ε, είναι εναρμονισμένοι. Δεν θα πρέπει τα οικονομικά και τα εμπορικά να υπονομεύουν την ανάπτυξη και τα πολιτικά. Γι' αυτό θα πρέπει να βάλουμε δεσμευτικέ ρήτρε και να εξασφαλίσουμε τη συνοχή των τριών πυλώνων. Έτσι ώστε όταν έχουμε ενδεχόμενη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει όποιος θίγεται να κάνει ε, καταγγελίες με τρόπο σωστό. Αυτό θα λένε τα Ηνωμένα Έθνη για τη σχέση με τις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να είναι δεδομένη σε όλους τους τομείς και να ενισχύεται σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η κοινωνία των πολιτών να εξισωθεί με τις επιχειρήσεις που το μόνο που τους νοιάζει είναι η κερδοφορία. Ενώ ο κόσμος ψάχνει την ε, αξιοπρέπειά του, τη ζωή του και καμιά φορά μόνο την επιβίωσή του. Θα πρέπει το εμπόριο που κάνουμε εμείς στο εσωτερικό αυτές σχέσεις να είναι δίκαιο, ε, βιώσιμο και στην υπηρεσία των πολιτών και όχι του κέρδους των συνήθων υπόπτων. Δεσμευτικά λοιπόν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η βιώσιμη ανάπτυξη και ρήτρε. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κοινωνικά στάνταρ και ε, περιβαλλοντικά και να έχουμε πάντα υπόψη την αηφορία και τη βιωσιμότητα του, του χρέους. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν υπέρ των πολιτών τους. Αλλιώς θα χάσουμε ξανά την ευκαιρία και θα πέσουμε στο συνήθι πατερναλισμό στις σχέσεις βορρά-νότου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. I been asked by any to have... Δεν μου ζήτησε κανένας άλλος το λόγο. Οπότε θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, Ματέο Γκογέτε. Θέλετε εσείς πρώτος να πάρετε το λόγο. Μετά από την, την ε, κρίση των φορών. Κούντουμσον λέγομαι. Από την ΤΕΦΚΟ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΤΕΒΕ και τον ε, βουλευτή Νόιζε για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς και για το σχέδιο έκθεσης καλωσορίζουμε την έκθεση πρώτα απ' όλα διότι ο, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το ζήτημα και καλός ο χρονισμός διότι ελπίζουμε σύντομα να δημοσιεύσουμε ε, την αξιολόγησή μας για τη Συμφωνία Κοτονού. Τις επόμενες μέρες προβλέπεται να δημοσιευθεί και θα δοθούν απαντήσεις σε κάποια από τα στήματα που έθεσε η κυρία Χόλμπρουκ. Ελπίζουμε το ταχύτερο δυνατό να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση αντικτύπου που διάφορα μελλοντικά σενάρια υπό το φως διαφόρων κριτήριων και ο Επίτροπος Μίντσα έχει πει ήδη και έχει εξηγήσει πως τον Νοέμβρη κατά πάσα πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει τις γραμμέ του μελλοντικές, ε, μελωδικούς προσανατολισμούς. Γι' αυτό σα λέω ότι είναι πολύ καλός ο χρονισμό διότι τροφοδοτείται η προϊόντα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι άλλο πολύ ενθαρρυντικό είναι πως βλέπουμε ε, τον ίδιο τρόπο σκέψης. Συγκλίνουν οι απόψεις μας και οπωσδήποτε αυτό συνιστά και ένα καλό εφαλτήριο. Ας περάσω στο περιεχόμενο τώρα. Χωρίς ακή, συμφωνία κοτονού δεν είναι απαραίτητα δημοφιλή ζητήματα, όμως η ουσία, οι σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ, σίγουρα αξίζει την προσοχή μας. Και όταν διαμορφώνουμε το μέλλον, όταν σχεδιάζουμε εκ νέου την πολιτική, χρειάζεται να σε εξέταση. Ιστορικά, αν το δούμε, άρχισε τη δεκαετία του 90 η διαπραγμάτευση για τη Συμφωνία Κοτονού, όμως παγκοσμίω ε, έχει αλλάξει άρδιν το σκηνικό. Η αλληλεξάρτηση είναι πολύ πιο έντονη. Ό,τι συμβαίνει και στην Αφρική κυρίως ε, μας επηρεάζει άμεσα στην Ευρώπη. Επίσης παγκόσμιες προκλήσεις, κλιματικές αλλαγές, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα υπερβαίνουν αυτές οι προκλήσεις στα σύνορα και δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε στα πλαίσια διμερών σχέσεων. Αρχίσαμε να εξετάζουμε τις σχέσεις μας με τις χώρες ΑΚΕ υπό το φως αυτών των νέων προκλήσεων. Τα συμπεράσματα δεν είναι σωστή λέξη γιατί ε, είναι τη γενέσιο η σκέψη μας. Θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το κεκτήμενο. Αυτές τις δεσμευτικές συμφωνίες των τελευταίων δεκαετιών να τις χρησιμοποιήσουμε. Μην χάσουμε αυτό το κεκτημένο όμως να επέλθει ουσιαστική αναβάθμιση. Πρώτα απ' όλα, κοινέ προτεραιότητες για τις παγκόσμιες προκλήσεις ταυτόχρονα να αποτυπωθεί το νέο ε, πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, στις συμφωνίες αυτές, ε, να αποτυπωθεί η Ευρωπαϊκή Συνένεση σε αυτές τις συμφωνίες, να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο προσέγγισης μας. Όπως ε, είπε και η Επιτροπή πις. Ε, ε, η ειρήνη, η δημοκρατία, η ευημερία και ούτω καθεξής, όπως είπατε και εσείς. Επίσης, να, να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι εταίροι μας. Γιατί υπερβαίνει το επίπεδο κυβερνήσεων η Συμφωνία Κοτονού. Κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικός τομέας, εθνικά κοινοβούλια ε, περιέχονται στη Συμφωνία ήδη. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την εταιρική σχέση. Τι γίνεται από πολιτικής πλευράς. Αυτό θα έχει κέρια σημασία. Πολιτικού τύπου διάλογο θα προωθήσουμε για να έχουμε απτά αποτελέσματα επί που Αυτό σημαίνει πως επιθυμούμε να διατηρήσουμε ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο, να διατηρήσουμε αυτή την διάσταση λαμβάνοντας όμως ε, περισσότερο την περιφερειακή διάσταση. Ε, ε, έχουν ενισχυθεί αυτές οι περιοχές, Καραϊβική, Ειρηνικό και κυρίως με την Αφρικανική Ένωση, αλλά και τα περιφερειακά μπλοκ, ΣΑΝΤΕΚ, Ένωση Νότιας Αφρικής, όλα αυτά τα περιφερειακά μπλοκ της Αφρικής είναι νέοι εταίροι και θα εφαρμόσουμε τη γνωστή σε όλους αρχή επικουρικότητας. και θα ανατεθούμε σε ποιο επίπεδο δεσμευσή θα κινηθούμε. Δηλαδή σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο υπήρου, σε επίπεδο χωρών και για να επιτύχουμε ε, τους στόχους μας όσους τις φιλοδοξίες που έχουμε. Αυτά από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε. Φαίνεται να, είμαστε, να υπάρχει ομοθυμία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κριστίνε Περόν τώρα παρακαλώ. Από πλευρά Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπατε και όντως συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ και με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ευχαριστήσω όμως τον κύριο Νόιζερ καθώς επίσης και του εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων που συνέβαλαν σε αυτή την πολύ επίκαιρη γνωμοδότηση. Να πω τα εξή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σαφώ να υπάρχει πολιτικό διάλογο, ιδιαίτερα προβεβλημένο αυτό και στι τροπολογίε και στην για την έκθεση. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τον πολιτικό αυτό διάλογο, το διάλογο επίση του άρθρου 8 και του άρθρου και τη διαδικασία του άρθρου 96. Ο πολιτικός διάλογος προβλέπεται στο άρθρο 8, όμως είναι πολύ πιο γενικός από αυτόν που έχουμε στα πλαίσια του άρθρου 96 και έχει σημειωθεί πρόοδο στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου τελευταία χρόνια. Πρέπει επίσης να σα ενημερώσω για το ότι λίγα χρόνια έχουμε ακόμα στη διάθεσή μα προτού προχωρήσουμε σε μια νέα μορφή σχέσεων με τις χώρες και Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μας αποθαρρύνει για τα όσα κάνουμε στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης έχουμε κάνει σημαντική προσπάθεια για να αξιολογήσουμε καταρχάς τι κάνουν τα κράτη-μέλη και αντιπροσωπείες μας στις ε, χώρες αυτές, ε, αν έχουν εξελογήσει το πολιτικό διάλογο, τι πηγαίνει καλά, τι επιδέχεται βελτιώσεις. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με το Συμβούλιο και με τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Λαμβάνουμε υπόψη μας και τη δημόσια διαβούλευση, στα πλαίσια της οποίας είδαμε ότι όντως θα πρέπει να εμπλέκεται περισσότερο η κοινωνία των πολιτών στον πολιτικό διάλογο και σε άλλους τομείς. Και θα υποβάλουμε κάποιες προτάσεις αυτή τη στιγμή ε, έχουμε συμφωνία επ' αυτών μετά τη διαβούλευση και συζητάμε ήδη από το θα συζητήσουμε από το φθινόπωρο και μετά με τα κράτη-μέλη για το πώς μπορούμε να κάνουμε τον πολιτικό διάλογο πιο αποτελεσματικό. Και θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ε, κάποια στιγμή αργότερα για το ζήτημα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση που θα πρέπει να έχουμε με επιμέρους περιφέρειες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η εξέλιξη των παγκόσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα και που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ως προς αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διατηρήσουμε ένα πολύ στενό διάλογο με τους εταίρους μας, με τις χώρες ΑΚΕ δηλαδή, ή ακόμα και με τις περιφερειακές συνιστώσεις των χώρων αυτών ή και με, το, ή και με τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκπονούμε εμεί συγκεκριμένε δεπτομερεί προτάσεις αν δεν προϋπάρχει ένας πολιτικός διάλογος με τις χώρες αυτές και αυτό ακριβώς είπε και ο Επίτροπος Μίμητσα πολλές φορές ότι όντως θα πρέπει να έχουμε πρώτη τη διαδικασία του διαλόγου προτού προχωρούμε σε διαπραγματεύσεις. Και κάτι ακόμα. Όταν πρόσφατα είχαν οι χώρες και τη δικιά τους τη σύνοδο, ένα από τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκε πολύ συχνά και στις συζητήσεις αλλά και στα έγγραφα, είναι ότι ε, πολλές χώρες ΑΚΕ ζητούν αναλογικότητα, επικουρικότητα και συμπληρωματικότητα. Τις αρχές δηλαδή αυτές να ληφθούν υπόψη στη μελλοντική σχέση που θα έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα ζητήματα συμπληρωματικότητα και ιδίω για την περιφερειακή αυτή συνεργασία και τη λεγόμενη προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να προκύψει από τη συνεργασία που έχουν χώρε αυτέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Νόζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ ξανά για τα σχόλια σας. Κοιτάξτε, Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή μας και το γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγάλη συναντήληψη είναι πάρα πολύ θετικό. Έχει αλλάξει η παγκόσμια κατάσταση και αλλάζει συνεχώς. Και ε, η θέση μας... Ε, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλαξε τελευταία στιγμή ε, λόγω και του Brexit. Σε μια έκθεση αυτό δεν μπαίνει τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα, αλλά μπορεί να γίνει. Ε, καλό θα ήταν την αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής να την είχαμε ήδη. Αλλά ακριβώ η σημερινή κατάσταση επιβάλλει να καταλήξουμε και χωρίς την αξιολόγηση σε μια κοινή στάση Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό φάνηκε από την προεργασία ε, για την έκθεση. Τα κράτη-μέλη ορισμένα έχουν πολύ επικριτική στάση. Και αν είμαστε στοιχημένοι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να βοηθήσουμε για τις μελλοντικέ σχέσεις ε, των χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πειράσουμε τα πράγματα. Να πω ξανά ότι καταρχήν και επί της ουσίας η εταιρική σχέση είναι σαφέστατο δικό μας αίτημα αυτό που θέλουμε είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, εταιρική σχέση, ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και ακούω ότι δεν θέλουν να περιμένουν, ε. Ε, αλλά ήδη από τώρα να μπουν ε, στον πολιτικό διάλογο, να μην περιμένουν τη διάδοχη συμφωνία, τόσο το καλύτερο και το ωραιότερο θα έλεγα. Άρα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που πετύχαμε. Τέλος θέλω να πω έτσι πάρα πολύ ε, κάτι που άκουσα στη συζήτηση. Αν η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ακόμα και η Ρωσία είχαν τέτοια συμφωνία τύπου κοτονού και θα την αξιοποιούσαν αλλά και θα τη συνέχιζαν. Uh, um, Ευχαριστώ. Έχουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ήδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη Γραμματεία ε, για την αποτελεσματικότητά της. 31 Αυγούστου θα ψηφίσουμε. Θα μας ενημερώσει η Γραμματεία. Άλλα δύο σημεία έχουμε. Ας περάσουμε ταχύτατα στο σημείο 10. Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλλιευτικών στόλων. Σχέδιο έκθεση για την σχέδιο χρηματοδότηση προς την Επιτροπή Αλληλείας για τον κανονισμό για την βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλληλευτικών στόλων. Η Μαρία Χολμπρουκ είναι η συγκητρία μας. Μαρία. Yeah, Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Για ποιο λόγο τώρα έχουμε επεξεργασία του κανονισμού η κοινή αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013 ε, αναθεωρήθηκε, έχει ειδικέ διατάξεις πλέον για τις εξωτερικές αλληλευτικές σχέσεις. Έχουμε εξωτερική αλληλευτική πολιτική. Ε, ε, βιώσιμη οικολογική διαχείριση ελευτικών πόρων. Από το έτος 2008 υπάρχει ένας κανονισμός για τα αλλιεύματα, για την αλλίευση. <laughs> Αλλά οι δραστηριότητες της Ένωσης, ελευτικές εκτός των δικών μας χωρικών υδάτων, θα πρέπει να βασίζονται στις ίδιες αρχές και αξίες ε, με εκείνη τη κοινή ελευτική πολιτική ε, στα ύδατα τη Ένωση. Θα πρέπει να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το στόλο τη, ανεξαρτήτω του που ελιεύει και ε, το τι γίνεται, να είναι σε θέση, λέω, να παρακολουθεί τι δραστηριότητε. Και άρα ο κανονισμό προβλέπει ε, αδειοδότηση αλίευση για αλευτικά σκάφη εξοκοινοτικά που δραστηριοποιούνται σε εξωτερικά χωρικά ύδατα ή εντός των δικών μας χωρικών υδάτων. Εδώ σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν διάφορες εξελίξεις ανάλογα με την κατάσταση και χρειάζεται να τις μελετήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσχώρησε στη διεθνή προσπάθεια του ΦΑΟ για την καταπολέμηση της ε, ε, παράνομης, αδήλωτης και λοιπά αλίας. Τώρα, για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά και τα κάνουμε. Ο κανονισμός του 2008 ίσχυε μόνο για ένα περιορισμένο τμήμα του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλλιεύει ε, στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ε, αποτέλεσμα ιδιωτικών συμφωνιών δεν το. Και όταν δεν υπήρχε τέτοια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κόσμος προχωρούσε σε ιδιωτικές συμφωνίες. Σημαίνει αυτό για την Αφρική, Μαδαγασκάρη, Τανζανία και Κένια. Επίσης δεν υπήρχαν ρυθμίσεις για ε, σκάφη που φέρουν κοινοτική σημαία, αλλά ε, που τα αναβλώνουν τύπου τσάρτερ για να πηγαίνουν να ψαρεύουν κάπου αλλού στο μέλλον αυτά όλα θα καλύπτουν ε, κάθε είδος αλίας και κάθε εργαλείο. Και ε, στα θετικά της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανήκουν τα εξής. Ε, ίσεις απαιτήσει και ρυθμίσεις για όλα τα σκάφη, τα αλλιευτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικά μας αλλιευτικά θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για να παίρνουν άδεια αλίες. Δύο σημαντικά κριτήρια ε, πρώτον, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να τους έχουν επιβληθεί βαριές κυρώσεις. Δηλαδή σκάφη ε, ε, που τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις διότι έχουν προβεί σε σοβαρές παραβάσεις και παραβιάσεις δεν παίρνουν άδεια. Η οδηγία θα πρέπει, μάλλον η αλία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και το κράτος σημαία, μάλλον οι πληροφορίε ε, για τη σημαία θα πρέπει να δίδονται από τον ιδιοκτήτη του σκάφου, από τον πλειοκτήτη δηλαδή και θα πρέπει να τεκμηριώνονται. Και όταν θέλουν κάποιοι να αλλιεύουν με ιδιωτικέ συμφωνίες θα πρέπει να φέρνουν ε, ανεξάρτητη επιστημονική μελέτη που να λέγει ότι αυτή η δραστηριότητα είναι η φόρος. Υπάρχουν περιορισμοί για το πώς μπορεί κανείς ως εξωτερική εταιρεία από τρίτη χώρα να αναβλώσει σκάφος με κοινοτική σημαία. Ε, επίσης, θα δημιουργηθεί μια τράπεζα δεδομένων δημόσια όπου θα αναγράφεται το όνομα του κάθε σκάφους και η σημαία που έχει, κάθε σκάφους που έχει άδεια αλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρχει ιδέουσα διαφάνεια είναι σημαντικό όλα τα ευρωπαϊκά αλλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για την αηφορία και στο εσωτερικό. Πόσο μάλλον που ο εξωτερικός μας αλλιευτικός στόλος υπόκειται στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει και αυτή να έχει τη δυνατότητα να κάνει καλύτερους ελέγχους. Με τη διαφάνεια λοιπόν και την δημόσια τράπεζα δεδομένων αυτό εξασφαλίζεται σε κάποιο βαθμό. Ο κανονικός θεσμός αυτός ε, αντιμετωπίζει το θέμα της παράνομης, αδήλωτης και ε, θέμετης αλίας και θα πρέπει να υποστηριχθεί. Υπάρχουν ε, ορισμένα ζητήματα δικονομίας που δεν έχουν οριμάσει και δεν έχουμε καταλήξει. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ επίγοντο θέμα και η πρωτοβουλία άριστη. Μερικές τροπολογίες από πλευράς μας είναι απαραίτητες, ωστόσο, για να βελτιώσουμε την έκθεση για τον κανονισμό. Το πρώτο είναι ο στόχος της αηφορίας. Προτείνεται για να υπάρχουν ε, συνεκτικές πολιτικές στην αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά δεν γίνεται σαφής αναφορά ε, το, στόχο, ε, στους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ κάναμε τροπολογίες συμπληρωματικά. Μετά υπάρχει η, η έννοια των α, αλλιευμάτων σε πλεόνασμα. Υπάρχουν τέτοια αλλιεύματα με βάση τον νέο κανονισμό. Τι σημαίνει αυτό. Ότι επιτρέπεται να ψαρεύονται συγκεκριμένα αλλιεύματα, αν θέλουμε να είμαστε βιώσιμοι, που δεν ψαρεύουν τα συγκεκριμένα κράτη, τα παράκτια, γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες τεχνικές. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε ε, να μην πηγαίνουμε εμείς με τα μεγάλα μας σκάφη να ψαρεύουμε αυτά που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι εκεί ε, με την παράκτη αλία και που ε, επεξεργάζονται σε κονσερβοποιήσεις που εργάζονται γυναίκες συνήθως. Και ένα τελευταίο έχει να κάνει με την αλλαγή σημαία. Ε, ορισμένα αλλιευτικά σκάφη έχουν μία σημαία ε, κάποιο διάστημα του έτους και μετά αλλάζουν σημαία ε, για να πάνε στα ίδια ύδατα και να συνεχίζουν να αλλιεύουν. Και μετά ξαναγυρνάνε στην προηγούμενη ευρωπαϊκή σημαία. Ωραία πράγματα. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός και μάλιστα ε, επιπλέον υπεραλίευση. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή προσπαθεί στον κανονισμό να το απαγορεύσει αυτό, αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Προς το παρόν να προβλέπουν πιο αυστηρούς κανόνες. Όταν αλλάζουν τη σημαία τους στα σκάφη μέσα σε 24 μήνες. Και ο περιορισμός είναι πάρα πολύ σύντομος. Αν έχετε ερωτήσει, είναι παρούσα και η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και μπορεί να απαντήσει πολύ καλύτερα από μένα σίγουρα τι λεπτομέρειε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I have... Uh, ε, ο κύριος Πόγκας και ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Μία διαδικαστική και μία άλλη για την ε, ουσία του ζητήματος. Σε επίπεδο διαδικασίας λυπάμαι διότι το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην αναπτυξιακή διάσταση. Αναφέρεται σε τεχνικά ζητήματα που είναι αρμοδιότητα, της αρμοδιότητας της Επιτροπής κατά τη γνώμη. Επίσης, είναι σημαντικό να τηρούμε τον εσωτερικό κανονισμό και να περιοριζόμαστε τις γνωμοδοτήσει μα στο πεδίο αρμοδιότητά μα. Πρώτη παρατήρηση επί τη διαδικασία. Δεύτερον, τη χάρη σε αυτό, στην αναθεώρηση του κανονισμού μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα τους εξωτερικούς αλλιευτικούς στόλους είτε στα πλαίσια των αλλιευτικών συμφωνιών ιδιωτικών ιδιών στα ανοιχτά ή και σε επίπεδο πόδα περιφερειακών οργανώσεων. Είναι πολύ καλή η πρόταση κανονισμού κάτι τη γνώμη μου. Επίσης, ε, αρμόζει να υπενθυμίσουμε την αρχή της συνεκτικότητας των πολιτικών σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο που εγκρίθηκε πέρυσι για την ανάπτυξη, δηλαδή ε, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Εγώ προσωπικά δύο τροπολογίες θα καταθέσω προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Φρανσούλικα. Έχουμε ένα καυτό ζήτημα για αύριο, γιατί έχει ψηφοφορία. Κυρίες και κύριοι, πρόεδρε. Ε, ε, κανονισμός 2006 του 2008. Αναθεωρείται αυτός ο κανονισμός ε, και πιστεύω ότι με την αναθεώρηση σε επίπεδο περιβάλλοντος, σε επίπεδο βιώσιμης αναπτύξης θα πρέπει να επιτύχουμε τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων. Η αναθεώρηση του κανονισμού για τις αδειοδοτήσεις είναι επιτακτική ανάγκη για να υλοποιήσουμε τους στόχους ελευθερικής μας πολιτικής και να επιτύχουμε την απλούστευση των τρέχουσων διατάξεων δεν μπορούμε να εντοπίσουμε όλα τα αλλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλλιεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ε, τρέχοντες κανόνες. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση για να υπάρχει υποπτία για τους εξωτερικούς αλλιευτικούς στόλους. οι διατάξει του τρέχοντος κανονισμού δεν επιτρέπουν αποτελεσματική και διαφανή υποπτία ε, και έλεγχο των ε, αλλιευτικών στόλων και αυτό μας οδηγεί σε ασάφεια και σύγκρουση αρμοδιοτήτων σε διάφορα επίπεδα επίπεδα ε, που εμπλέκονται στη διαδικασία. Υπάρχουν επίσης ε, ελλείψεις ως προς διατάξεις. Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις δεν θα μπορέσουμε με βιώσιμο τρόπο να διατηρήσουμε τους ελευτικούς πόρους και θα πληγεί η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να το αποφύγουμε. Ο προτινόμενος κανονισμός πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να έχει θετική, θετικό αντίκτυπο στις τρίτες χώρες που δίνουν αυτές τις άδειες στα δικά μας αλληλευτικά σκάφη. Βελτιώνοντας τις επιδόσεις των εξωτερικών αλληλευτικών στόλων θα μπορέσουμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα σε ε, παγκόσμιο επίπεδο για τη διαχείριση των αλληλευτικών πόρων και κάποιες τρίτες χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο τον νέο κανονισμό για να τροποποιήσουν το δικό του σύστημα και να εφαρμόσουν τον έλεγχό του ε, για σκάφη που ε, είναι εγώ έχω τη δική του σημαία. Σας ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση. Μήπω πρέπει να την απευθύνουμε στην Επιτροπή, μάλλον, όχι στην κυρία Χολιμπροκ. Εγώ δεν είμαι ειδικό για αυτό το κανονισμό. Αλλά αναρωτιέμαι, τι γίνεται με το προσωπικό στου εξωτερικού ελευθερικούς στόλου, με τα πληρώματα. Έχουμε Ε, ακούσει διάφορα για τα σκάφη που φέρουν τη σημεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλιεύουν εκτός, ότι δεν καλύπτονται από το εργατικό δίκαιο τη εργασιακής διατάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι τους εκμεταλλεύονται του τους ανθρώπους. Ποιος κανονισμός ε, είναι εφαρμοστέος. Ε, ξέρω ότι εσείς τα έχετε εξετάσει αυτά τα ζητήματα και στο παρελθόν. Ναι, ναι, ε, σόκαρε επίση το ότι έμαθα ότι αυτοί που δουλεύουν και στα φέρει μπότ ορισμένε φορέ δεν καλύπτονται από τι εργασιακές διατάξει. Υπάρχουν ε, ε, Ε, μπορείτε να μας πείτε ακριβώς ε, τι ισχύει και αν ασχολείται κανείς με αυτό το ζήτημα. είναι θέμα χρηματοδότηση, γιατί σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα. Για να ακούσουμε την Επιτροπή. Η κυρία... Η κυρία Αμάντο, για την DG Ο... Ποιο, ποιος θέλει το πρώτο στο λόγο. DG Μάρε. Ευχαριστώ, Άννα Όλιβερτα, από την DG Μάρε. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχά για τη γνωμοδότησή σας αυτή. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον συντάκτη της γνωμοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι όντω η γνωμοδότηση αυτή συμβάλλει πολύ στην όλη διαδικασία έγκριση ε, τη ε, πρότασης αυτή για την βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών ηλεκτρικών στόλων. Με την άδειά σα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σα πω πω έχουν τα πράγματα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με την πρόταση αυτή και στη συνέχεια θα μπορούσα να απαντήσω και στο δικό σας το ερώτημα, κυρία Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, στις 15 Φεβρουαρίου λέβε χώρα ένα συμβούλιο όπου οι υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της πρότασης αυτής αλλά εξέφρασαν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με το επιπλέον διοικητικό άκθος που μπορεί να επιφέρει η πρόταση αυτή, καθώς επίσης και σε σχέση με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας αδειοδότησης. Από το Φεβρουάριο λοιπόν μέχρι σήμερα εργαζόμαστε σε έξι διαφορετικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε το κείμενο, να το καταστήσουμε πιο απλό, να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής να καταφέρουμε να κάνουμε την πρόταση αυτή να συνάδει περισσότερο με το βασικό κανονισμό όσον αφορά την αλία. Η πρόταση αυτή έχει να κάνει με την βιώσιμη αλία, αλλά έχει να κάνει και με την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας και έχει να κάνει βασικά με την υποπτία και τον έλεγχο των ελευτικών σκαφών μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ελεύουν δηλαδή σε ύδατα τρίτων χωρών. Επεξεργαζόμαστε λοιπόν το κείμενο αυτό με τη βοήθεια τη Προεδρία και με του επιτετραμένου των κρατών μελών σε θέματα τελεία προκειμένου να βελτιωθεί σε τεχνικό επίπεδο. Έχουμε καταφέρει επίση να μειώσουμε τον πολύ μεγάλο ρυθμό δεδομένων που απαιτούσαμε. Ξέρετε ότι υπήρχαν δύο παραρτήματα που απαιτούσαν δεδομένα για παντό είδου δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή συνδέσαμε το κείμενο αυτό με άλλα κείμενα τα οποία έχουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθετικά και ουσιαστικά χρησιμοποιούμε δεδομένα τα οποία ήδη υφίστανται σε άλλες βάσεις δεδομένων. Επομένως, οι υποχρεώσεις υποβολής δεδομένων και το όλο το διοικητικό έργο που πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο έχουν απλουστευθεί πάρα πολύ ενώ παράλληλα, παράλληλα με συγχωρείτε, διατηρούμε τις βασικές αρχές και τους βασικούς στόχους της σημαντικής αυτής πρότασης. Στις 15 Ιουνίου έγινε μια συνεδρίαση της Κορεπέρα και εκεί οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών και η Προεδρία τάχθηκαν υπέρ των βελτιώσεων που έχουμε επιφέρει στο κείμενο και μάλιστα η Προεδρία έστειλε και μία επιστολή στο Συμβούλιο ζητώντας την έγκριση γενικής προσέγγισης βάσει του συμβαστικού κειμένου του Συμβουλίου της Προεδρίας και μάλιστα επετεύχθη μια συμφωνία στην, στο Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα τα κράτη-μέλη τάχθηκαν σαφώς υπέρ των βελτιώσεων που είχαμε επιφέρει στο κείμενο. Έχουν απλουστευτεί λοιπόν και έχουν εναρμονιστεί όλες οι διαδικασίες όπως σας είπα, ζητάμε πολύ λιγότερα δεδομένα πλέον. Η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στο παρελθόν παρουσίαζε μία επικάλυψη με άλλες διεθνείς αλλιευτικές συμφωνίες ή σε, οι ανάλογες υποχρώσεις υπήρχαν στα πλαίσια άλλων διεθνών ελευτικών συμφωνιών. Αυτή τη στιγμή οι επιπλέον υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων είναι απλώς συμπληρωματικέ. Σε καμία περίπτωση δεν συμπίπτουν, δεν επικαλύπτουν οι φυστάμενες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Και έχουμε συμπεριλάβει και κάποιες νέες διατάξεις στην πρόταση αυτή, προκειμένου να ρυθμίσουμε ένα ζήτημα το οποίο ήδη υφίστατο στην πρόταση εξ αρχής, δεν είναι αρκετά σαφές. Είπαμε ότι χρειαζόταν ένα νέο τμήμα, ένα νέο κεφάλαιο για τις λεγόμενες βόρειες συμφωνίες. Δηλαδή, να καταφέρουμε να ρυθμίσουμε καλύτερα την αλίευση σε ύδατα όπου αλλιεύουν και άλλες χώρες όπως η Νορβηγία και άλλες σκανδιναβικές βόρειες χώρες. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Το Συμβούλιο συμφώνησε για μια γενική προσέγγιση. και έχουν ξεκινήσει βέβαια και οι συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή Ελίας. και μετά το καλοκαίρι θα μας σε θέση να δούμε και την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Να απαντήσω τώρα στην ερώτησή σας και να κάνω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις που νομίζω ότι θα πρέπει να κάνω τώρα στα πλαίσια αυτής της συζήτησης. Όσον αφορά αυτά που είπε και η περίοδος των 24 μηνών. Κοιτάξτε, η πρόταση αυτή ευθυγραμμίζεται με το βασικό κανονισμό. Έχουμε ένα νέο βασικό κανονισμό για την αλία που εγκρίθηκε πριν από δύο περίπου χρόνια και στον κανονισμό αυτό έχουμε το άρθρο 31, σημείο 9 συγκεκριμένα, που αναφέρεται ακριβώς ε, στο ζήτημα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Προβλέπεται λοιπόν αυτή η χρονική περίοδος των 24 μηνών. Στα πλαίσια λοιπόν του κανονισμού αυτού προσπαθήσαμε να εναρμονίσουμε την πρόταση αυτή με τους ήδη φυστάμενους κανόνες, προκειμένου να υπάρχει απόλυτη συνέπεια και συνεκτικότητα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να επαναλάβουμε εδώ πέρα αυτή την περίοδο των 24 μηνών όσον αφορά τους ελέγχους συμμόρφωσης. Και βέβαια Υπάρχουν ορισμένε χώρε οι οποίε είχαν θέσει χαμηλότερε απαιτήσει όσον αφορά το ζήτημα αυτό τη βιωσιμότητα. Στην πρόταση αυτή υπάρχουν γενικά κριτήρια επιλεξιμότητα, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα σκάφη τα οποία επιθυμούν να αλλιεύσουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου λοιπόν να αλλιεύσει ένα ευρωπαϊκό σκάφο εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να έχει άδεια αλλίας και η άδεια αυτή αλεία μπορεί να δοθεί από τα κράτη-μέλη μόνο αν πληρούνται τα κριτήρια αυτά επιλεξιμότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και αυστηρό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό τα σκάφη αυτά να μην έχουν κάνει σημαντικές παραβάσεις, να έχουν συγκεκριμένο αριθμό μητρώου, να μην έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Θεωρούμε λοιπόν το κείμενο δίνει τις κατάλληλες διασφαλίσεις, τα κατάλληλα εχέγγυα για την αδειοδότηση των σκαφών αυτών. Απαντήσω λοιπόν και στο δικό σας ερώτημα, κυρία Πρόεδρε, τα εργασιακά δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα στους κοινοτικού αυτούς στόλους. Ξέρετε ότι τα σκάφη αυτά τα οποία φέρουν κοινοτική σημαία θα πρέπει να συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Πρέπει να συμμορφώνονται λοιπόν με το δίκαιο αυτό. Και κάθε κράτος μέλος ε, σημαίας θα πρέπει να ελέγχει ότι όντως υφίστανται τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία ισχύουν και σε εθνικό επίπεδο, ότι όντως αυτά εφαρμόζονται στα πλαίσια του εν λόγω σκάφους. Δεν ξέρω, άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, ήταν μακρός και λύση εξηγήσει. Ο κ. Κνότ, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, ΔΕΦΚΟ. Εκπροσωπώ σήμερα εδώ αυτή τη Γενική Διευθύνση να μην μακρηγορήσω, γιατί ε, η καθήλυνα αρμόδια είναι η DGMAR. Εμείς ε, είμαστε συνδεδεμένοι γενική διεύθυνση και ακούσατε τώρα τη συνάδελφο που τοποθετήθηκε. Θέλω μόνο να τονίσω πώς ε, συμμορφούνται ο κανονισμός αυτός με την αναπτυξιακή πολιτική. Συμβάλλει, δεν είναι μόνο συμβατό, συμβάλλει στην αναπτυξιακή πολιτική ε, ως προς ε, μια σειρά ε, στοιχείων που θα υποστηρίξουμε για να προωθήσουμε την αναπτυξιακή πολιτική. Πολύ σας ευχαριστούμε. Ναι, θα σε σχέση με προηγούμενα καθεστώτα σίγουρα στην βελτίωση. Θέλεις να προσθέσεις τίποτα Μαρία. Σε παρακαλώ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Για τον κύριο Πόνγκα. εσείς μιλήσατε για συνεκτική πολιτική η ελευτική πολιτική συνδέεται άρρηκτα με την αναπτυξιακή πολιτική, οπότε μπορούμε να το δούμε κάπως ευρύτερα ε, και να το κοιτάξουμε και από κάποια δική μας σκοπιά της Επιτροπής Ανάπτυξης. Thank you very much, colleague. Deadline for amendments is... Ευχαριστώ. Προθεσμία για τις τροπολογίες Τετάρτη 13 Ιουλίου, 12. Η ώρα το μεσημέρι. Τελευταίο σημείο, 11. Συμφωνίες τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τα την κουκ. ΚΟΚ. Ε, ο κύριος Πόγκα είναι ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ. Σύντομα θα σας παρουσιάσω αυτό το σχέδιο συμφωνίας ε, και το πρωτόκολλο για αλληλευτικά ζητήματα με τα νησιά Κούκο. Στον ελληνικό είναι αυτά. 40 ε, τράτες, ε, κυρίως ισπανικές, ε, θα μπορέσουν να λιεύουν τόνο κοντά σε αυτά τα νησιά για τέσσερα έτη ανανεώσιμη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει 735.000 τα δύο πρώτα χρόνια και 700.000 τα επόμενα δύο. 350.000 ετησίω για την υποστήριξη ε, της ανάπτυξης του αλευτικού τομέα ε, στα νησιά Κουκ. Ε, υπερβαίνει αυτό το κονδύλι σε σχέση με το 11ο ΦΕΝΤ. Επίσης έχουμε τα δικαιώματα πρόσβασης που θα πληρώνουν οι πλειοκτήτες. Πολύ καλή συμφωνία τηρούνται όλα τα κριτήρια της νέας αλληλευτικής πολιτικής, κυρίως για τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων, για την επίθυνη και βιώσιμη αλληλεία και την τήρηση, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της πρόθεση της διαφάνειας. Επίσης είναι σημαντική η συμφωνία διότι χάρη σε αυτή Μπορεί να προωθηθούν οι αρχέ τη βιώσιμη αλληλεία στον ελληνικό από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ζητώ να δώσετε την κατάθεσή σα για να ε, συναυθεί αυτή η συμφωνία. Ευχαριστούμε. Ξεκάθαρη, ξεκάθαρη η έκθεσή σα, ξεκάθαρη και οι συστάσει σα. Ο κύριο Φραντσούλικα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας ε, θα ήθελα, αν μου το επιτρέπετε, να υποστηρίξω τη θέση του εισηγητή, φυσικά θα υπερψηφίσω. Θα υπάρχουν θετικέ επιπτώσει για τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων, για τη βιώσιμη αλεία, για την καταπολέμηση τη άναρχη λαθρέα και παράνομη αλεία θα προωθηθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ε, η δημοσιονομική συνεισφορά αντιστοιχεί σε υποστήριξη πολιτικής για τη ε, διαχείριση των αλλιευτικών πόρων και τη στήριξη του εγχώριου αλλιευτικού τομέα στα νησιά Κουκ. Ε, Μαρία, θέλεις το, το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ, Μωρίς Πόγκα. συμφωνώ Digimare, DigiDevco, έχετε... Ε, εσείς είσατε κατά βάση αρμόδια. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πόγκα. Το σχέδιο εκθεσής του μπορούμε πλήρως να σας υποστηρίξουμε. Ήθελα μόνο να τονίσω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι νέες βιώσιμες συμφωνίες, αλληλευτικές συμφωνίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνεται πρόσβαση ε, στους αλληλευτικούς μας τόλους ε, νέα ύδατα, αυξάνει την παραγωγικότητα και οι αλληλευτικές δυνατότητες ε, διατηρούνται στην περιοχή, διότι ξέρουμε όλοι ότι η εξέπνευση η συμφωνία στον Ειρηνικό, η προηγούμενη συμφωνία στον Ειρηνικό και πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας στην περιοχή. Ε, ως προς και την ε, Περιφερειακή Επιτροπή για το Κεντρικό Κοινό του Ειρηνικό. Δεν εκπροσωπευόμαστε πλέον ως ο κράτος, καταλαβαίνετε, οπότε ε, ούτε και ως αλλιεύων κράτος. Οπότε θα ενισχυθεί η θέση μας. Αυτό ήθελα να τονίσω. Κατά τα συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Ευχαριστούμε την Τζιντεύκο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Όπως είπε και ο κύριος Πόγκα, τα ποσά τα οποία προβλέπονται εδώ πέρα είναι υψηλότερα από το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή θέση και να καταφέρουμε κατά επέκταση να υποστηρίξουμε έτσι τη νήσου Κουκ, πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πόγκα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι, όλα ήταν σαφή. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. 14 Ιουλίου 5η το μεσημέρι είναι η ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών. 31 Αυγούστου θα ψηφίσουμε. Ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνεδρίαση. Θα συνεδριάσουμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί και ξεκινάμε με ψηφοφορίες. Παρακαλώ πολύ φέρτε την κάρτα.